morning. Καλή σας μέρα. Ας ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συνεδρίαση. Θα αρχίσω να μιλάω Ιταλικά, ως συνήθως. Προτιμώ να προεδρεύσω στα Ιταλικά. Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης, την έγκριση της ημερησίας διάταξης. Τα πιο σημαντικά θέματα που θα συζητήσουμε σήμερα αφορούν τις αναφορές για ρήπανση στο Τάραντο, ε, χρηματοδότηση του γεωργικού τομέα στην Ιρλανδία. Αποστολές στη Δανία, Ελλάδα, κάλυψη, υγειονομική κάλυψη των Βρετανών πολιτών στην Γαλλία, διαβίβαση διοικητικών εγγράφων στην Πολωνία και πρωτοβουλίες, ε, πρωτοβουλίες ε, για προληπτικές εξετάσεις ε, πριν από τη γέννηση. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ένας συναλφος δεν μπορεί να έρθει στις εργασίες της Επιτροπής μας γιατί είχε ένα δυστύχημα, όχι μεγάλο. Είναι στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Δεν θα συμμετάσχει στις εργασίες. Θα έχουμε και κάποιες αλλαγές στη μερική διάταξη. Κυρίως ε, τις ψηφοφορίες και τις συζητήσεις για τις ε, προτάσεις ε, για αποστολές που θα ξεκινήσουν στις 11 και όχι το απόγευμα. Και για την αποστολή στη Γαλλικία, η αποστολή που θα γινόταν τον Νοέμβριο αναβλήθηκε. Το 8 ε, το ζήτησε ο συντάκτης να ακυρωθεί και το σημείο 19 επίσης ακυρώνεται γιατί οι συντονιστές δεν μας είπαν ποιος θα είναι ο εισηγητής. Στο σημείο 5 θα πάρει το λόγο όχι ο κ. Πάξας, αλλά ο κύριος Μπιτζότο και τα σημεία 6, 9, 7 και 11 θα είναι παρόντες οι συντάκτες. Για τις συνεδρίες των συντονιστών θα ξεκινήσουμε 11 και 45. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, θεωρώ ότι έχει κάποια διάταξη. Δεν βλέπω να έχετε αντιρρήσεις. Ο κύριος Αλαβράκος. Καλημέρα σα, καλημέρα του συναδέλφου, Δεν έχω αντιρρήσει, αλλά επειδή επιγόντω πρέπει να φύγω για την Αθήνα, θα ήθελα να κάνω κάποιε σύντομε δηλώσει που θα ήθελα να κατεχωρηθούν στα πρακτικά. Πρώτον, στη συζήτηση του σημείου 6 της ημιλησία διάταξη για την αναφορά τη κυρία ε, Μπιζότο, σχετικά με την παραβίαση του δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι ΡΑΗ, σα γνωστοποιώ την υποστήριξη τη ομάδα μα ώστε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή. Στο σημείο 11 της ημιλησίας διάταξης ε, δίδω τη θετική μου ψήφο για την έγκριση της έκθεσης σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στη Δανία. Και τρίτον, υπενθυμίζω τη στήριξή μου στο κοινό κείμενο το οποίο απέστειλε ο κύριος Γιάρ εκ μέρους της ομάδας μου, του Άλντε, του S&D και του ΕΛΚ για τις μεθόδους εργασίας της Επιτροπής Αναφορών που θα συζητήσετε στη συνάντηση των συντονιστών. Τέλος, για τη διερευνητική έκθεση στην Πολωνία συντάσσομαι με τον εισηγητή. Και παρακαλώ να εγκριθεί σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σαλαβράκο. Κύριε Μπούλαντ, αν θα φύγετε κι εσείς όπως και ο κύριος Σαλαβράκος, ε, να είστε σύντομα. Αλλιώς, ε, στο σημείο 4 να πάρετε το λόγο, στα διάφορα. Οκ, okay, προχωρώ τότε. Θέλω να εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδρίασης της 16ης. Τι θέλετε για την ημερήσια διάταξη, να πάρετε το λόγο, παρακαλώ. Eh, Καλημέρα. Εγώ προσωπικά Εκ μέρους όμως του Κριστέλου θα σα προτείνω για την έκθεση σχετικά με την Πολωνία αν μπορούμε να αναβάλουμε την ψηφοφορία για μια προσεχή συνεδρία τη Επιτροπή μα. Ενημέρωσα τον κύριο Τέιλορ γραπτό για αυτό το θέμα. Χθε το βράδυ μου είχε διατυπωθεί το αίτημα, πολύ αργά, πολύ καθυστερημένα, και ζήτησα από τι ομάδε τη γνώμη του. ε, οι δύο ομάδε είναι αντίθετε. Και τώρα ο κύριο Αλαβράκος. Άρα αναγκαστικά πρέπει να κάνω την ψηφοφορία αυτή, γιατί είχε γραφτεί στην ημερήσια διάταξη. Πάω στο δεύτερο σημείο, έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 16 η και 17 η Σεπτεμβρίου. Αντιρρήσεις. με τα πρακτικά όσο έχουν. Ξέρετε ότι μετά μια πρώτη, αφού διανεμηθεί η ημερήσια διάταξη, με τις αποφάσεις που έχουν κληθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των συντονιστών και που είναι το κείμενο που μόλις ψηφίσαμε, δεν συμπεριλαμβάνει τις αποφάσεις των συντονιστών. Γιατί? ούτως ή άλλως αυτές δεν διαβάζονται όπως γίνεται συνήθως, αλλά σήμερα το απόγευμα θα διαβαστούν παρόλα αυτά. Ε, μαζί με τις αποφάσεις που θα πάρουν σήμερα οι συντονιστές στις 11.45. Επομένως αυτές οι αποφάσεις θα γίνουν εκτελεστές μετά την ψηφοφορία της Επιτροπής. Για τις επιπλέον ανακοινώσει του Προέδρου, που αφορούν το παράρτημα Β. Ξέρω ότι, ξέρετε μάλλον ότι πρέπει να κάνετε παρατηρήσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω για αυτό το θέμα. Ο κ. Μπουλάντ όμως μου ζήτησε το λόγο για τα διάφορα. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να επενθυμίσω ότι η αναφορά 900 79 για τον κύριο Ζήρου ε, θα παρακαλέσω να μείνει ανοιχτή διότι δημοσιοποιήθηκε η υπόθεσή του στη Γαλλία, εκδόθηκε ε, από τη Γερμανία στη Γαλλία και από την, ε, το ανάποδο μάλλον. Και γι' αυτό σας παρακαλώ να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά στα σημεία Β, θα ήθελα να λάβω το λόγο και να ε, μιλήσω για αυτή την πρόταση. Κοιτάξτε, για να είναι όλα ξεκάθαρα, οι παρατηρήσεις για το σημείο Β της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζονται γραπτός στην Πρόεδρο και η Πρόεδρος ανακοι... διαβάζει αυτές τις παρεμβάσεις. Έτσι δεν χρειάζεται κάθε πρόβλημα να το συζητάμε ιδιαιτέρως. Τέλο πάντων, το αίτημα του κύριου Μπουλάν πάντω το κατέγραψε η γραμματεία. Ο κύριο Γκόμε. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σα παρακαλέσω να μην κλείσετε δύο αναφορέ. Την 1998 του 12 η οποία αφορά τη διπλή των Σλοβάκων υπηκόων. Όταν το συζητήσαμε το Μάιο Ξέραμε ότι έπρεπε να αναμένουμε την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου τότε, που όμως δεν έχει προβεί στην ετοιμιγωρία του ακόμα. Θα ήθελα λοιπόν να περιμένουμε την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου και να μην κλείσουμε πριν από αυτήν ε, την εν λόγω αναφορά. Είναι θέμα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Για άτομα τα οποία παίρνοντα δεύτερη υπηκότητα χάνουν κάποια άλλα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη δεύτερη αναφορά, την 1571 του 12 για λόγω αναφορά προέρχεται από γκροϊπικό που έχασε τα στεξιδοτικά της δικαιώματα γιατί δεν είχε αρκετό χρόνο να προετοιμαστεί Υπήρχαν και πολλέ άλλε παρόμοιε αναφορέ. Εμεί ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη για τι επτώσει τη κρίση σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη, για να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να βάλουμε αυτή την καταγγελία ε, μαζί με άλλες που προέρχονται και από την Ουγγαρία και άλλα από άλλες χώρες. Ευχαριστώ κύριε Γκόμες. Εντάξει, κατάγραψαμε το έτοιμά σας. Θα το λάβουμε υπόψη. στη συνάντηση των συντονιστών. Και τα δύο αιτήματα θα τα λάβουμε υπόψη στη συνάντηση των συντονιστών. Συνεχίζουμε με την μέση διάταξη. Φτάσαμε στο σημείο 5. Νομοδότηση για την 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο τη εφαρμογή του δικαίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω σας είχα προαναγγείλει, θα πάρει το λόγο η κυρία Μπιτζότο. Ή ο κύριο Μπιτζότο μάλλον. Αντί για τον κύριο Πάξα. Θα διαβάσω τι μου είπε, μια και δεν μπορούσε να έρθει με το πρωί. Η 21 η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μιλάνε γενικά για τις ε, ευρωπαϊκές οδηγίες και την εσωμάτωσή τους. Ε, μιλάμε για οδηγίες ε, στατιστικών ε, και υποτίθεται ότι είναι δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το 2011 ε, βελτιώθηκαν τα νομοθετικά κείμενα της, των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν παραβιάσεις που δείχνουν ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα ενσωμάτωσης που πρέπει να επιληθούν. Η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα εφαρμογής του, Ευρωπαϊκού, ε, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα διάφορα κράτη-μέλη διαφέρει από κράτος σε κράτος, ανάλογα με τους τρόπους εφαρμογής που έχει ε, επιλέξει κάθε κράτος μέλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει ε, να λάβει υπόψη τι αρχέ τη επικουρικότητα και τη αναλογικότητα. Ε, οι νομοθετικέ πράξει τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι αποτελεσματικέ και να δίνουν ε, με το μικρότερο δυνατό κόστο το μεγαλύτερο όφελο. Η Κομισιόν θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην εφαρμογή του δικαίου και του δικαιώματο του κάθε πολίτη να υποβάλει αιτήσει. Αναφορές και για την δικαίωμά του και να αναγνωρίζονται αμέσως οι περιπτώσεις παραβιάσεων. Θα πρέπει πάντα η Κομισιόν να ενημερώνει την Επιτροπή Αναφορών με ενδελεχείς έρευνες, στατιστικές κτλ. Μετά από αναλύσεις που κάνει η ίδια η Κομισιόν. Είναι, είναι αναγκαίο να βελτιώσουμε τις... την συνεργασία μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων, ε, Ευρωκοινοβουλίου, Είναι ανάγκη να βελτιώσουμε την, ανάγκη, την συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων, ε, Εθνικών Κυβερνήσεων και Ευρωκοινοβουλίου. Ούτως ώστε η μεταφορά των κοινοτικών νομοθετικών πράξεων στο Εθνικό Δίκαιο να είναι απόλυτα διαφανής. Είναι απαραίτητο επίσης να μειώσουμε το γραφειοκρατικό άχθος και διοικητικό άχθος. Η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει μία λεπτομερή αξιολόγηση των επιπτώσεων και των πλεονεκτημάτων κάθε νομοθετικού κειμένου, ούτω ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα των, της απόκρισης των κρατών μελών. Ευχαριστώ κύριε Μπιτζότο. Είναι μια πρώτη σκέψη, ένας πρώτος προβληματισμός για την έκθεση. 30 Οκτωβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών στις 5 το απόγευμα. Οι τροπολογίες θα εξεταστούν και θα ψηφιστούν στις 26 Ενδεκάτου, 26 Νοεμβρίου. Θέλει κάποιο το λόγο. Από την άποψή μας ε, χρήση βελτίωση στο κείμενο, χρειάζονται και τροποποίησει. Μας δώσατε την προθεσμία, οπότε μέχρι να λήξει θα καταθέσουμε και εμείς τις δικές μας τροπολογίες για να βελτιώσουμε αυτό το κείμενο, ώστε να προσεγγίσει τις δικές μας προσδοκίες. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Ε, υπάρχει εκπρόσωπος της Κομισιόν που θέλει να πάρει το λόγο. Τώρα. Παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ε, ευχαριστώ πολύ για το πρώτο αυτό σχέδιο προτάσεων. Θα ήθελα να κάνω τις εξής πρώτες παρατηρήσεις από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα εκτιμούσαμε ο ρόλος ε, των αναφορών ε, στις διαδικασίες παράβασης ε, να αναγνωρίζεται και θα ήθελα να αναφέρω ότι στην ετήσια έκθεση στο βασικό έγγραφο υπάρχει ειδικό τμήμα αφιερωμένο αποκλειστικά στις αναφορές που λάβαμε το 2011 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις δράσεις που έχει αναλάβει η Επιτροπή πάνω στις αναφορές αυτές. Και επίσης, αν κοιτάξετε το δεύτερο τμήμα, θα δείτε την ε, λεπτομερή ανάλυση ανατομέα πολιτικής. Σε κάποιους από τους τομείς ε, πολιτικής υπάρχουν κοινοβουλευτικές δραστηριότητες. Εάν λοιπόν η Κομισιόν ε, λαμβάνει αναφορές Αυτές αναφέρονται ανά τομέα πολιτικής και θα θέλαμε να διατηρήσουμε την πρακτική αυτή και στο μέλλον. Δεύτερον, αναφέρατε τη μείωση του διοικητικού άχθους και την ε, πιο αποτελεσματική νομοθεσία. Το πρόγραμμα REFIT της Κομισιόν ε, στοχεύει ακριβώς σε αυτό και έχουμε και ένα πρόγραμμα μείωσης του γραφειοκρατικού άχθους για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ε, όταν συμμορφώνονται με κανονισμούς και άλλους κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούσαμε και παρατηρήσεις και πρόταση ότι μπορεί τα κράτη-μέλη να χρειαστούν κάποια βοήθεια στην μεταφορά του κοινοτικού δικαίου ε, ή ε, ότι μπορεί να χρειάζεται βοήθεια κατά την αλλαγή κυβέρνησης σε εποχές εκλογών. Η εφαρμογή του ε, δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κυρίως υποχρέωση της διοίκησης των κρατών μελών και η δυνατότητά μας να βοηθήσουμε είναι περιορισμένη και εξαρτάται και από την δική τους αποδοχή. Πάντως ε, θα είναι πολιτική της Κομισιόν να στηρίζουμε οδηγίες με σχέδια εφαρμογής που να βοηθούν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν στην πράξη πιο αποτελεσματικά τις διατάξεις ε, των οδηγιών. Θα ήθελα να σχολιάσω το πρόγραμμα EU Pilot. Δεν αποτελεί μηχανισμό παραπώνων. Έχουμε λάβει εκκλήσεις από διάφορες ε, επιτροπές, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αντικαταστήσουμε το ρυθμιστικό υπόβαθρο του EU Pilot με ε, κάτι που να έχει νομικά δεσμευτική μορφή. Θα ήθελα να σημειώσω ότι η δημιουργία του συστήματος EU Pilot βασίζεται σε διμερείς ρυθμίσεις ανάμεσα στην Κομισιόν και τα κράτη-μέλη. Η αντικατάσταση της βάσης αυτής με ένα νομικά δεσμευτικό μέσο Ε, για να το πω ήπια θα είναι μονομερής τροποποίηση ε, της παρούσας δομής του EU Pilot. Εάν υπήρχε κανονισμός ή πρόταση, θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας ότι τα κράτη-μέλη δεν θα καταπιούν πολύ εύκολα την αντικατάσταση αυτή της νομικής βάσης. Αυτή πάντως είναι η δική μας εκτίμηση. Και τέλος, στο σημείο 17 έγινε πρόταση τα κράτη-μέλη να καταβάλουν προσπάθειες για την ολοκλήρωση διαδικασιών παράβασης προτού φτάσουν στο δικαστήριο. Πράγματι είναι πολύ δύσκολο να δίνουμε πληροφορίες σχετικά με ε, τις ε, ε, κλειστές διαδικασίες παράβασης, διότι δεν ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τον τύπο και το κοινό. Αλλά οι κανόνες διαφάνειας για τις περιπτώσεις που έχουν κλείσει είναι πολύ πιο χαλαροί σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν για τις εκκρεμούσες υποθέσεις. Και αν κάποιος θέλει να ελέγξει αν η Κομισιόν έκλεισε μια υπόθεση λόγω πλήρους συμμόρφωσης ενός κράτους μέλους. Αυτό είναι απολύτως δυνατό να γίνει. Με ε, έτοιμα πρόσβαση στα έγγραφα. Ευχαριστώ. So uh, uh, Ευχαριστώ. Μπορούμε να κλείσουμε το θέμα αυτό και να προχωρήσουμε. Σημείο 6. Αναφορά από την Μάρα Μπιτζότο, Τζίνο Ατζέρντε, Ροζάριο Μποσκέρι, εξ ονόματος της Επιτροπής Λίπερα Informazione της ραδιοτηλεόρασης, με μια αρχική παρουσίαση 11.432 υπογραφών, ε, στις οποίες προσθέθηκαν και άλλες 3.000 μέχρι χθες το βράδυ. Η αναφορά αφορά τη σύγκρουση που υπάρχει ανάμεσα στον τρόπο διαχείρισης της ΡΑΗ και, την, ε, το ευρωπαϊκό δίκαιο. Έχουμε παρόντες τους ε, εκπροσώπους της Επιτροπής αυτής, της Επιτροπής ε, Libera Informazione και έχουμε και τον κύριο Μποσκέρη που είναι ο δεύτερος συντάκτης της αναφοράς αυτής, στον οποίο δίνω το λόγο. Καλημέρα σας κύριε Ευρωβουλευτές. Είμαστε εκπρόσωποι της Επιτροπής Κομιτάτο Λίμπερα Informazione Λίμπερα Τελεβιζίδα. Ε, εκπροσωπούμε 55.000 ανθρώπους και επί 30 χρόνια είμαστε ενεργοί σε όλη την ε, επικράτεια της Ιταλίας. Ε, με ένα στόχο. Θέλουμε να καταργηθεί το τέλος υπέρ της ΡΑΗ, ούτως ώστε όλοι οι πολίτες ε, της ε, Ιταλίας να έχουν μια ανεξάρτητη και πλουραλιστική ενημέρωση. Στην Ιταλία υπάρχουν τόσες ε, οργανώσεις και επιτροπές όπως η δική μας. Και όλοι μας ε, έχουμε, δίνουμε μία ε, κοινή μάχη ελευθερίας και πολιτισμού για να καταργήσουμε ένα φόρο ο οποίος είναι απόλυτα άδικος και άνισος, που είναι το τέλος υπέρ της ΡΑΗ. Ξεκίνησε αυτός ο φόρος να επιβάλλεται από το 1938, επί φασιστικού καθεστώτος. Ο, το τέλος υπέρ της ΡΑΗ είναι από τους πιο άδικους φόρους στην Ιταλία. Γιατί η ΡΑΗ δεν είναι δημόσια τηλεόραση. Στην πραγματικότητα είναι στα χέρια των κομμάτων και χαρακτηρίζεται από μία δραστηριότητα χωρίς, χωρίς πλουραλισμό, ανεξαρτησία και διαφάνεια της πληροφορίας. Μην ξεχνάμε τις ε, άπειρες περιπτώσεις προβληματικών ε, ζητημάτων με τη ΡΑΗ που την καθιστούν απόλυτα προβληματική. Παρά το γεγονός ότι εκατομμύρια Ιταλοί πληρώνουν το τέλος της ΡΑΗ, παρά τα άπειρα έσοδα που έχουν από τις διαφημίσεις στη ΡΑΗ, παρά τη δημόσια χρηματοδότηση από το Ιταλικό κράτος, η ΡΑΗ κάθε χρόνο έχει απίστευτες τρύπες του προπολογισμό της. Το 2012 το deficit, ο... δηλαδή το έλλειμμα της ΡΑΗ ήταν 245 εκατομμύρια ευρώ λόγω της κακοδιαχείρισης της ΡΑΗ. Όλα αυτά ποιος θα πληρώνει συνεχεία, ο Ιταλός φορολογούμενος. Ευχαριστώ. Θέλω να δώσω το λόγο στον δικηγόρο τον κύριο Ρίο, ο οποίος μας βοηθάει σε αυτή τη μάχη που δίνουμε. Ευχαριστώ. Καλημέρα Πρόεδρε. Κύριοι Ευρωβουλευτές, η αναφορά δείχνει ότι ο Ιταλικός νόμος, ο οποίος υποχρεώνει τους Ιταλούς πολίτες να πληρώνουν το, το τέλος αυτό, έρχεται σε απόλυτη αντίφαση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επανέρχομαι, γιατί ε, δεν δόθηκε απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα αιτήματά μας. Καταρχάς, το Ιταλικό δίκαιο παραβιάζει το θεμελιώδες δικαίωμα ισότητας και ενημέρωσης των πολιτών. Για να μην πληρώνουμε, πληρώνει το Τέλος, ο Ιταλός πολίτης είναι υποχρεωμένος μέσω μιας απίστευτα δύσκολης διαδικασίας, βυζαντινής θα έλεγα διαδικασίας, να ε, παρετηθεί από τη χρήση της τηλεόρασής του, που πρέπει να μπει μέσα σε ένα σάκο και να τον σφραγίσει ένας ε, δημόσιος υπάλληλος. Ουσιαστικά δηλαδή παρετείται από την τηλεόρασή του ο Ιταλός πρέπει να την καταλήψει και του στερείται το βασικό μέσο πρόσβασης στην πληροφόρηση από, όλους τους, από όλα τα κανάλια εθνικά και ξένα. Ακόμα και αν πει ότι εγώ μόνο από τη ΡΑΗ θέλω να παρατηθώ και όχι από τα υπόλοιπα κανάλια. Αυτό το γεγονός παραβιάζει το, το θεμελιώδες δικαίωμα ελευθερίας και έκφρασης που α, καταγράφεται στο άρθρο 11 της Χάρτας Ευρωπαϊκής Ένωσης και που δίνει το δικαίωμα στον ε, Ευρωπαίο πολίτη ε, να λαμβάνει πληροφορίε, να ενημερώνεται χωρίς ξένες παρεμβάσεις. Η ΡΑΗ ισχυρίζεται ότι οι χρηματοδοτήσεις που λαμβάνει με το τέλος δεν παραβιάζουν την ε, νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις και δεν παραβιάζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό από τη στιγμή που δίνει ε, παρέχει δημόσια υπηρεσία. Η ΡΑΗ όμως ε, όλο και πιο συχνά παραβιάζει τις, τους όρους της ε, σύμβασής της που της επιτρέπουν να εισπράττει το, το τέλος όπως το αποδεικνύει εδώ και 30 χρόνια το κανάλι ΡΑΗ ΣΑΤ. Το το Συμβούλιο Επικρατείας της Ιταλίας ε, με την απόφαση 4336 του 2013 καταδίκασε τη ΡΑΗ γιατί χρησιμοποίησε με απαράδεκτο τρόπο τα έσοδα που λαμβάνει από το τέλος ε, και αυτό το, λέει το ανώτατο δικαστικό σώμα της Ιταλίας. Επίσης, η ΡΑΗ παραβίασε τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και άλλες σοβαρές παρατυπίες που αφορούν την, το σήμα της ΡΑΗ. Η ΡΑΗ έχει μία άδεια για αυτό το σήμα και έχει την συμβατική υποχρέωση να εξασφαλίσει την καθολικότητα της δημόσιας αυτής υπηρεσίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 2 εκατομμύρια περίπου Ιταλοί που δεν λαμβάνουν το σήμα της ΡΑΗ, δεν, το... φτάνει ως αυτούς. Αυτό σημαίνει ακόμα μια μεγάλη βαθιά ε, διάκριση ανάμεσα στους πολίτες. Ανάμεσα σε αυτούς που, μπορούν, που λαμβάνουν το σήμα της ΡΑΗ και αυτούς που δεν το λαμβάνουν, όχι λόγω του ότι δεν θέλουν, αλλά λόγω της ευθύνη της ΡΑΗ. Και ακόμα πιο σοβαρό, η ΡΑΗ βάζει αυτούς τους ανθρώπους, ακόμα και αυτούς, να πληρώσουν το τέλος για μια υπηρεσία που δεν έχουν λάβει ποτέ και ε, δεν πρόκειται να λάβουν. Καμία απόφαση σε καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καμία νομοθεσία δεν μπορεί να επιβάλλει την ε, πληρωμή μιας υπηρεσίας η οποία δεν δίδεται. Ακόμα πιο επιβαρυντικό στην περίπτωσή μας είναι ότι η ΡΑΗ ήξερε από την αρχή ότι δεν πρόκειται να δώσει σε αυτούς τους πολίτες αυτού του είδους την υπηρεσία. Αν αυτός ο θεμελιώδης και βασικός κανόνας πληρώνω μόνο εφόσον μου δίδεται η υπηρεσία ισχύει γενικά για τους πολίτες, προφανώς θα πρέπει να ισχύει και για, τις, ε, κρατικές, ε, για τους κρατικούς φορείς, όπως η ΡΑΗ, που είναι υποχρεωμένοι μέσω σύμβασης να ε, παράσχουν υπηρεσία προς το κοινό συμφέρον, αλλά που δεν το κάνουν όμως και παρόλα αυτά εισπράττουν από όλο τον κόσμο. Ζητάμε λοιπόν η Επιτροπή σας, η Κομισιόν μάλλον, να ξαναδεί την θέση αυτή, να δει την κατάσταση και να αναγνωρίσει τις καταφανείς παραβιάσεις της ΡΑΗ και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Μην, ξεχνάμε, μην ξεχνάτε επίσης ότι πέρα από τις υπογραφές που μαζέψαμε έχουμε άλλες 3.100 υπογραφές ε, που μαζεύτηκαν τελευταία. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαρτορέλη θέλει το λόγο για να απαντήσει, ε, να μιλήσει μάλλον εξ ονόματος της ΡΑΗ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Η δημόσια τηλεόραση στην Ευρώπη υποβαλόταν σε ειδικέ ρυθμίσεις, γιατί είναι αναμφίβολο και αναγνωρίζεται ο ρόλος που παίζει η δημόσια τηλεόραση σε, σε τις κοινωνίες μας, που είναι δημοκρατικές, ε, πολύμορφες, ε, πλουραλιστικές κτλ. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με αυτούς τους στόχους. Υπάρχει κρατική χρηματοδότηση της ε, δημόσιας τηλεόρασης, τηλεόρασης και αυτό ε, επιβεβαιώθηκε στο πρωτόκολλο του Άμσταρντα του, της 2 Οκτωβρίου του, του 1997, όπου λέγεται ότι τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για να αποφασίσουν για τον τρόπο χρηματοδότησης της δημόσιας τηλεόρασης. Ο τρόπος ε, που λειτουργεί η δημόσια τηλεόραση επομένως, ε, ρυθμίζεται από τα κράτη-μέλη. Με βάση το ρόλο που παίζει η δημόσια τηλεόραση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εκφραστεί σε ό,τι αφορά τα θέματα του τέλους υπέρ της ΡΑΗ για την Ιταλία, μετά από εκθέσεις και παρουσιάσεις που είχαν να παρουσιαστεί στο παρελθόν από εμπορικές τηλεοράσεις στην Ιταλία και η Κομισιόν έδωσε μία απάντηση πολύ πλήρη τον Οκτώβριο του 2003 και τον Απρίλιο του 2004, δύο αποφάσεις, όπου επιβεβαιώθηκε οριστικά η απόλυτη συμβατότητα του τέλους υπέρ της ΡΑΗ με τους κανόνες ε, για τις ε, κρατικές ενισχύσεις ε, των δημοσίων φορέων. Επίσης, η Κομισιόν συμφωνεί με τον ορισμό της δημόσιας υπηρεσίας που είχαν δώσει οι Ιταλικές αρχές και δεν εμφανίστηκε πουθενά ε, προφανές λάθος από πλευράς ΡΑΗ. Υπάρχει απόλυτη αναλογικότητα της ε, χρηματοδότησης της ΡΑΗ σε σχέση με την ε, υπηρεσία που προσφέρει η ΡΑΗ. Δεν υπάρχει καθόλου υπερβολική ε, πληρωμή, η πληροβολική αποζημίωση της ΡΑΗ για τις δημόσια υπηρεσία που προσφέρει. Η ανακοίνωση του 2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ της δημόσιας τηλεόρασης είναι και αυτή μια σημαντική απόφαση. Έχουν ενσωματωθεί εκεί και οι διάφορες αποφάσεις των δικαστηρίων, καθώς και η διαβόητη απόφαση που αναφέρει η αναφορά και αναφέρεται ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν απόφαση, που προσφέρουν υπηρεσία δημόσια, ε, χρηματοδοτούνται χωρίς αυτό να θεωρείται κρατική ενίσχυση. Η ανακοίνωση επίσης υπενθυμίζει αυτό που έλεγε και το πρωτόκολλο του Άμστερνταμ, ότι είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών να διαλέξουν τον μηχανισμό που θα εξασφαλίσει την ε, εποπτεία και τον τρόπο άσκησης των, ε, της, ε, της υπηρεσίας αυτής. Αν υπάρχει πρόβλημα θα πρέπει να υπάρξουν διορθωτικά μέτρα. Στην Ιταλία όπως ξέρουμε δημιουργήθηκε ένας φορέας, η GCOM, για την για τις τηλεπικοινωνίες. Είναι ένας ανεξάρτητος και αυτόνομος μηχανισμός και που θέλει, θα πρέπει να εξασφαλίσει τη σωστή, το σωστό ανταγωνισμό όλων των φορέων και την ελευθερία των Ιταλών πολιτών. Επίσης, τη δημόσια υπηρεσία στον τομέα της της τηλεόρασης την προσφέρει η ΡΑΗ. Αυτό το αποφασίζει επίσης ο ίδιος φορέας. Η ΡΑΗ επίσης έχει χωριστά λογιστικά βιβλία για τα τέλη που εισπράττει από τους Ιταλούς πολίτες για την παροχή αυτής της δημόσιας υπηρεσίας. Και υπάρχει ε, ένα σχήμα, ένα σύστημα που ε, που έφτιαξε αυτός ο φορέας, η GCOM, ε, που το στέλνει στο Υπουργείο το αρμόδιο και ελέγχεται από μία ανεξάρτητη αρχή στο τέλος. Ε, επαληθεύονται λοιπόν όλες οι παράμετροι και το κατά πόσον είναι ικανοποιημένοι οι χρήστες. Όπως, λένε, όπως λέει η σύμβαση της ΡΑΗ, η GCOM στην ετήσια έκθεση του 2013 επιβεβαίωσε ότι η ΡΑΗ χρησιμοποίησε την ε, χρηματοδότηση από το τέλος για την υλοποίηση της ε, υπηρεσίας της αυτής, δηλαδή την παροχή δημόσιας υπηρεσίας, ε, σεβόμενη όλες τις ε, διατάξεις της σύμβασής της και ποιοτικά και ποσοτικά. Αυτό πιστοποιήθηκε από την ετήσια έκθεση της GCOM και επιπλέον επαναλαμβάνεται ότι υπάρχει αυτό το χωριστό σύστημα λογιστικών βιβλίων που προβλέπεται στη ΡΑΗ και υπάρχει και υποχρέωση δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της όλων των ετησίων λογαριασμών που πιστοποιούνται από την ε, ελεγκτική εταιρεία. Επίσης στο site ε, ε, δημοσιεύονται διάφορα προγράμματα που χρηματοδοτεί το τέλος. Σε ό,τι αφορά τα σημεία που μόλις ακούσαμε από τους συντάκτες της αναφοράς, η λήψη του σήματος που για μας είναι σημαντική, ε, για αυτήν τι έχουμε ξεκινήσει. Από το 2008 ε, η ΡΑΗ έχει ξεκινήσει τη διαδικασία μετατροπής του σήματος σε ψηφιακό σήμα με βάση τους τρόπους που προβλέπει το Υπουργείο Οικονομικών και με βάση τα όσα προβλέπει η σύμβασή μας. Ε, όμως αυτή η σύμβαση δεν κάνει συγκεκριμένη αναφορά σε περιοχές της Ιταλίας και σε συγκεκριμένες κοινότητες, αλλά ε, μιλάει για ποσοστά κάλυψης της Ιταλικής επικράτειας σε σχέση με αυτά τα ποσοστά κάλυψης, εφαρμόσαμε σωστά τα όσα προβλέπει η σύμβαση με βάση τις υποχρεώσεις ε, που μας είχαν επιβληθεί. Είναι αλήθεια ότι με σκοπό να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την, ε, τη λήψη του σήματος, πώς θα για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα ε, λο, κάνουμε ό,τι μπορούμε χρησιμοποιώντας το multiplex 1 ε, προκειμένου να μην υπάρχουν ε, προβλήματα ανάμεσα στα διάφορα σήματα των διαφόρων α, καναλιών. ΡΑΙ 1, ΡΑΙ 2, ΡΑΙ 3. Ούτως ώστε να ξανασχεδιάσουμε, να ξανακατανείμουμε τις συχνότητες ανάμεσα στα διάφορα κανάλια. Ζητάμε λοιπόν από την Επιτροπή Αναφορών να ακυρώσει, να μην δεχτεί τα επιχειρήματα της αναφοράς και να μη δεχτεί να ανοίξει παραβίαση, να ανοίξει διαδικασία για παραβίαση εις βάρος της ΡΑΗ, γιατί έχουμε σεβαστεί όλες τις υποχρεώσεις και τη σύμβασης και χρησιμοποιούμε τα έσοδα από το τέλος όπως πρέπει. Ούτε θέλουμε επίσης να καταργηθεί το τέλος αυτό, γιατί το τέλος το πληρώνει μόνο όποιος έχει συσκευή τηλεοπτική. Αυτά, Πρόεδρε, ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Πίκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα τέλη τηλεόραση δεν είναι δημοφιλή σε κανένα κράτος μέλος. Υπάρχουν πολίτες σε πολλά κράτη μέλη που μας στέλνουν επιστολές να καταργηθούν αυτά τα τέλη. Η απάντησή μας είναι πάντα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο αποτελούν τα τέλη μια δυνατότητα ε, των κρατών μελών για το πώς θα οργανώσουν την ε, χρηματοδότηση ε, της δημόσιας τηλεόρασης. Λαμβανωμένου υπόψη του πρωτοκόλλου που προσταθήκε στην συνθήκη του Άμστερνταμ πέρα από τους κανόνες της Κομισιόν. Τα κράτη-μέλη λοιπόν καθορίζουν τα τέλη ανάλογα με το αν υπάρχει τηλεόραση ή όχι, αλλά κράτη-μέλη λένε ότι κάθε νοικοκυριό θα πρέπει να πληρώνει άσχετα από το αν ο κόσμο βλεπει βλέπει τηλεόραση ή όχι. Αλλά κράτη-μέλη έχουν αποφασίσει να το κάνουν αυτό με διαφορετικό τρόπο, στις κάτω χώρε, για παράδειγμα. Έχουν καταργηθεί τα τέλη. Ε, πληρώνεται, από πληρώνεται από τα φορολογικά έσοδα η δημόσια τηλεόραση. Ε, αυτό πάντω αποτελεί επιλογή των κρατών μελών. Μπορώ να επιβεβαιώσω αυτά που είπε η εκπρόσωπο της ΡΑΗ σχετικά με το γεγονός ότι η Κομισιόν στο παρελθόν έχει εξετάσει το θέμα των κρατικών ενισχύσεων προ τη ΡΑΗ και διαπίστωσε μετά από κάποιες ε, τροπολογίες ε, των Ιταλικών αρχών ότι είναι απολύτως συμβατό το σύστημα και δεν είδα τίποτα στην αναφορά που να με κάνει να έχω αμφιβολίες σχετικά με το αν θα πρέπει να επανεξεταστεί η αναφορά αυτή. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Εάν οι αναφέροντες λένε ότι η ΡΑΗ δεν συμμορφώνεται με την εντολή της ε, περί δημόσιας υπηρεσίας ε, σε διάφορα σημεία, ε, εάν διαπιστωθεί παράβαση δηλαδή, αυτό δείχνει ότι υπάρχει σύστημα εποπτείας και ότι αυτό το σύστημα λειτουργεί. Εάν η ΡΑΗ δεν συμμορφώνεται, επιβάλλεται πρόστιμο, επιβάλλεται κάποια κύρωση. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου με τον τρόπο που θα έπρεπε να υπάρχει και ε, τέτοιο που ζητάμε από όλα τα κράτη-μέλη να έχουν. Και φαίνεται να λειτουργεί. Κυρία Πρόεδρε, λοιπόν, η θέση μας είναι ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη να ξεκινήσει νέα έρευνα της χρηματοδότησης της ΡΑΗ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξεκινάει η συζήτηση. Κυρία Μπιτζότα, πρώτη και καλύτερη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το τέλος της ΡΑΗ είναι ένας χώρος που μισούν οι Ιταλοί γιατί είναι άδικος. Δεν θέλουν οι Ιταλοί πολίτες να πληρώσουν το τέλος της ΡΑΗ γιατί η ΡΑΗ δεν είναι ε, δημόσια τηλεόραση και δεν προσφέρει δημόσια υπηρεσία. Είναι μια απαράδεκτη ανομαλία που είναι αδικαιολόγητη. Ούτε στη δημόσια φύση της ΡΑΗ, ούτε στα προγράμματα της τηλεόρασης αυτής. Ο δικηγόρος που μίλησε πριν έθεσε κάποια θέματα τα οποία θα ήθελα να υπογραμμίσω ακόμα μια φορά. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για δημόσια τηλεόραση, γιατί η ΡΑΗ δεν εξασφαλίζει ε, την υπηρεσία αυτή σε όλους τους πολίτες που πληρώνουν το τέλος. Μεταξύ των εγγράφων που σας δώσαμε στο φάκελο θα βρείτε την καταγγελία και άλλων ε, οργανώσεων πολιτών ε, που έκανε μάλιστα και ομαδική αγωγή κατά της ΡΑΗ, γιατί οι πολίτες δεν λαμβάνουν το σήμα της ΡΑΗ, δεν πιάνουν τη ΡΑΗ. Μιλάμε για δημάρχους διαφόρων ε, περιφερειών ε, και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για να ελέγχουν αυτές τις υπηρεσίες. Αλλά υπάρχουν όμως και καταγγελίες βουλευτών. Υπάρχουν τουλάχιστον 2 εκατομμύρια άτομα, όπως μας λένε, που δεν λαμβάνουν το σήμα της ΡΑΕ και παρόλα αυτά πρέπει να πληρώσουν το τέλος. Εν συνεχεία. Δεν είναι δημόσια τηλεόραση αυτή η δημόσια υπηρεσία, γιατί όπως καταγγέλουν οι εθνικές ε, οργανώσεις για την προστασία και τη βοήθεια των ε, πολιτών, το να πληρώνει κανείς το τέλος χωρίς να λαμβάνει τις υπηρεσίες είναι απόλυτη διάκριση. Επομένως, θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτές οι επιστολές, κυρία Πρόεδρε, αξίζει να διαβαστούν. Γιατί υπάρχουν δύο σημαντικές οργανώσεις που στηρίζουν αυτή την αναφορά, γιατί πάρα πολλά άτομα στην Ιταλία κάθε μέρα δεν έχουν το δικαίωμα πρόσβαση στην πληροφορία και σε μεγάλο μέρος προγραμμάτων της ΡΑΗ. Ελάχιστα είναι τα προγραμμάτα της ΡΑΗ, να μην πω δεν υπάρχουν, που η Επιτροπή Αναφορών νομίζω πρέπει να παρέμβει γιατί μεταξύ των, είναι μεταξύ των υπεύθυνων φορέων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλάει για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες κτλ. Επίσης η απόφαση του Αυγούστου του 2013 από το Συμβούλιο Επικρατείας της Ιταλίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν νομίζω ότι την είδε την απόφαση αυτή, γιατί αλλιώ θα έχει απαντήσει διαφορετικά. Είναι μια αποφάση που καταδικάζει την ΡΑΗ και την ΑΤΖΙΚΟΜ, που είναι η, δημόσ... εθνική αρχή, που είναι η αρχή που πρέπει να επαγρυπνεί και να εποπτεύει τη ΡΑΗ. Καταδικάστηκε για σοβαρότερε παραβιάσει των υποχρεώσεων παροχή δημόσιας υπηρεσία. γιατί η ΡΑΗ δεν επιτρέπει σε διαφόρους πολίτες ε, παρά μόνο να έχουν πρόσβαση στην ε, πλατφόρμα TV SAT ε, και τους αποκλεί από διάφορα προγράμματα. Επομένως, τα χρήματα από το τέλος χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που δεν είναι δημόσια υπηρεσία. Οι αποφάσεις της... Οι απαντήσεις που μας δίνει η Επιτροπή είναι γελίες μας αναφέρει αποφάση του 2003 και 2005 που δεν είχαμε περάσει από την αναλογική ψηφιακή τηλεόραση που έγινε το 2009 στην Ιταλία. Όμως η Κομισιόν δεν αναφέρει την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας του Αυγούστου του 2013 που λέει το εξή και παρακαλώ τον εκπρόσωπο της Επιτροπής να, να ακούσει. Δημιουργώντας την πλατφόρμα TVUSAT, ε, η, ΡΑΗ δεν σέβεται την, ε, τον, ε, τους ίσους όρου με τους οποίου πρέπει να παίζει η ΡΑΗ με τους υπόλοιπου ε, ιδιωτικούς φορείς. Πρόκειται, επομένως, η, τα άρθρα 107 και 108 της ε, Συνθήκης λειτουργία Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάζονται γιατί ε, δεν υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Ε, και υπάρχουν προβλήματα με τις ε, κρατικές ενισχύσεις. Ε, δεν γνωρίζετε αυτές τις αποφάσεις ε, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι μετά από την απόφαση η Κομισιόν θα πρέπει να παρέμβει και να ξεκινήσει μια διαδικασία επιπαραβάση κατά τη ΡΑΙ και κατά τη Ιταλία. Γιατί η απόφαση καταδικάζει και την Τζικόμ, που είναι η υπηρεσία η οποία θα πρέπει να εποπτεύει την δημόσια ραδιοτηλεόραση. Ζητώ λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξανασκεφτεί την απόφασή τη και να αλλάξει γνώμη και να ξεκινήσει μια έρευνα για τη σωστή χρήση τη δημόσια χρηματοδότηση από πλευρά ΡΑΙ η Κομισιόν μετά από αυτές τις νέες πληροφορίες θα πρέπει να αποφασίσει αν η ΡΑΗ είναι ακόμα δημόσια τηλεόραση και αν γι' αυτό η ΡΑΗ δικαιούται να, λαμβάνει το, να εισπράττει το τέλος. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσει μια διαδικασία επί παραβάση Κομισιόν κατά της ΡΑΗ λόγω, των, λόγω της παραβίασης των κανόνων α, ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Επίσης, ε, απαντήστε Κομισιόν για το σημείο 20 της ε, αναφοράς. Στην ε, Ιταλία, ένας Ιταλός πολίτης, με βάση ένα νόμο του 1938 του φασιστικού καθεστώτος, μπορεί να αρνηθεί να πληρώσει το τέλος. Ε, σε αυτή την περίπτωση όμως του σφραγίζεται η συσκευή της τηλεόρασής του. Ε, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συσκευή του. Ε, την κλείνουν σε έναν σάκο και σφραγίζεται. Ο πολίτης επομένω δεν μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες όπως προβλέπει το άρθρο 11 του χάρτη για τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωση. Δεν μπορεί επομένω, μια και δεν έχει τηλεόραση του η οποία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πια, να παρακολουθήσει καμία εκπομπή, ε, κανένα δελτίο ειδήσεων, ούτε στα Ιταλικά, ούτε, από, ούτε σε καμία άλλη γλώσσα από άλλο κανάλι. Γιατί η Κομισιόν δεν λέει τίποτα για αυτό το σημείο. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Η ΡΑΗ δεν εγγυάται την ελευθερία πληροφόρησης και τον πλουραλισμό. Η ΡΑΗ ανήκει στα κόμματα. Ε, οι διορισμοί γίνονται από τους πολιτικού. από τους πολιτικούς. Επομένως, δεν υπάρχει πληροφόρηση ελεύθερη και ανεξάρτητη. Δεκάδες πράγματα, δεκάδες παραδείγματα μπορούμε να φέρουμε, αλλά σας λέμε τα τελευταία. Ρώμη, 11 Οκτωβρίου, ε, δήλωση του Διευθυντή της ΡΑΗ. Αυτά τα χρόνια η εικόνα της δημόσιας τηλεόρασης στην Ιταλία, αλλά όχι μόνο, ε, στυλιτεύτηκε λόγω ε, πολύ στενών σχέσεων με την πολιτική. Υπάρχει πρόβλημα με την αμεροληψία της. Ο ίδιος δηλαδή παραδέχεται ότι ε, τα κάνει πλάκα και με τους πολιτικούς. Ρώμη 30 Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος ε, επαγρύπνησης της ΡΑΗ, που είναι μια ειδική επιτροπή που εποπτεύει τη δημόσια τηλεόραση, Παρακαλώ πρέπει να κλείσετε. Έκανε κατάληψη στην, στα γραφεία της ΡΑΗ για να καταγγείλει τα, τις τρύπες στον προπολογισμό. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όμως. Και κλείνω. Η καταγγελία του Κόντα που είναι μια Ιταλική οργάνωση πολιτών, που καταγγέλνουν ότι πληρώνονται κάτι απίστευτα ποσά τα στελέχη της ΡΑΗ. Ε, δύο εκατομμύρια πληρώνεται ένας παρουσιαστής της ΡΑΗ. Σε αυτό νομίζω θα μιλήσουν και οι συνάδελφοι. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά το θέμα της ΡΑΗ και να εκφράσει μια γνωμοδότηση με βάση παρατηρήσεις που ακούσατε. Νομίζουμε ότι η καταγγελία που έχει αναφορά ε, και όλα τα στοιχεία που ακούσατε σήμερα είναι μόνο ένα ελάχιστο τμήμα του προβλήματο. Νομίζω όλα αυτά θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω. Να δοθεί η ιδιαίτερη προσοχή από την Επιτροπή Αναφορών. Τα προβλήματα των χρηστών. Ε, τα προβλήματα που αναφέρουν όλοι αυτοί οι δήμαρχοι. Δεν μπορεί όλα αυτά να τα περάσουμε στον τούκου. Το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν θα πρέπει να παρέμβουν και συμπερασματικά ζητάω από την Επιτροπή Αναφορών, από την Πρόεδρο Ματσόνη να προγραμματίσω μια συνάντηση με την Επιτροπή Εποπτείας της ΡΑΗ και ζητάω από την ε, Επιτροπή, την Κομισιόν, να κάνει μια σοβαρή εξέταση όλων των προβλημάτων που ακούσατε σήμερα. Η γνωμοδότηση που σας δώσαμε είναι πολύ σοβαρή και τεχνηριωμένη. Η δική σας είναι ε, μεροληπτική, ελλειπής και γελία. Ο κ. Μοτζέσκι. από το, Ευρωπαϊ... από το Βελγικό Κοινοβούλιο, από, την... Ε, από το... και μάλιστα από την Επιτροπή Αναφορών του Βελγικού Κοινοβουλίου. Και τώρα ο κύριος Μποστινάρου. Θα μιλήσω ρουμάνικα, Πρόεδρε. Câteva constatări și voi spune Θα ήθελα να πω ευθύς εξ αρχής ότι είμαι ένθρωμος οπαδός της δημόσιας τηλεόρασης. Είμαι πεπισμένος για το ρόλο και τη σημασία της δημόσιας τηλεόρασης στην ευρωπαϊκή κοινωνία, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την επίθεση ε, τηλεόρασης ε, που θα τη χαρακτήριζα υποκουλτούρα και που είναι προσβλητική πολλές φορές και σίγουρα υπάρχουν ε, πολλά ιδιωτικά συμφέροντα στην τηλεόραση με Απογοήτευσε πάντως ε, πάρα πολύ η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά το τέλος τηλεόρασης, αυτό πράγματι υπάρχει στα περισσότερα κράτη-μέλη. Ωστόσο, από τη Μάγνα Κάρτα και μετά οποιοδήποτε φόρος, οποιοδήποτε τέλος πρέπει να βασίζεται σε μια κοινωνική σύμβαση. Πληρώνω ένα φόρο, πληρώνω ένα τέλος σε αντάλλαγμα για την ε, παροχή μιας υπηρεσίας. Εκατομμύρια όμως Ιταλοί πολίτες, ναι μεν υποχρεούνται να πληρώσουν το τέλος στη ΡΑΕ, αλλά δεν παίρνουν κανένα αντάλλαγμα, δεν παίρνουν κάποια υπηρεσία ως αντάλλαγμα. Αυτό δεν ενοχλεί καθόλου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών. Μα δεν έχουμε ακόμα μια οδηγία που αφορά την προστασία των καταναλωτών αξιότιμη εκπρόσωπη της Κομισιόν. Εσείς μάλλον την ξεχνάτε ή κάνετε σαν να μην υπάρχει αυτή η οδηγία. Δεύτερον, αυτό το τέλος έγινε ε, υποχρεωτικό με την έννοια ότι όλοι οι πολίτες του κράτους μέλους υποχρεούνται να έχουν μια σύμβαση παροχής υπηρεσίας χωρίς να την έχουν ζητήσει όμως. Εντάξει, σε μια δικτατορία ίσως ε, επιβάλλει κάποιος να δεχθείς κάτι που δεν θέλεις, αλλά σε μια δημοκρατική ε, κοινωνία, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, αυτό δεν είναι δυνατόν. Ούτε και στη Ρουμανία, στη χώρα μου, Αξιότιμε εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν έχουμε την επιβολή αυτή από ε, κάποιο πάροχο υπηρεσίας. Δηλαδή, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, θέλετε να δείτε ή να μην δείτε τηλεόραση, θα πληρώσετε. Μα τι είναι αυτό. Αυτό είναι παράλογο στην ε, Ρουμανία το άνατο το δικαστήριο ξεκάθαρα δήλωσε ότι αν κάποιος δεν θέλει να του παρέχεται η υπηρεσία αυτή, δεν υποχρεώται να την πληρώνει. Και από ό,τι γνωρίζω, η ρουμανική, η ρουμανική νομοθεσία εμπνέεται από το αρχαίο ρωμαϊκό δίκαιο μέσω του Ναπολεόντιου κώδικα, αλλά τέλος πάντων. Τι να πω, τρίτο σημείο. Μιλάμε για κατάφορη ε, κατάφορο περιορισμό που αντιβαίνει σε όλη την ομολογία του Δικαστήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Διότι, εάν σε ένα κράτος μέλος ε, που η τηλεόραση πρέπει να θεωρείται ιδιωτική περιουσία ε, του κάθε ανθρώπου, η τηλεόραση, το μηχάνημα αυτό που έχει σπίτι σου, είναι ιδιωτική προσωπή, είναι περιουσία και μόνο με απόφαση δικαστήριου μπορεί να κατασχεθεί. Από τον Απολέοντα ισχύει αυτό. Δεν υπήρχε τηλεόραση βέβαια τότε. Δεν ξέρω, μπορεί να θέλετε να δώσετε την ευλογία σας για μια διαφορετική λύση, αλλά για να σφραγιστεί, να κατασχεθεί μια τηλεόραση χρειάζεται απόφαση δικαστηρίου, απόφαση δικαστή. Αλλιώς εγώ που είμαι ο κάτοχος, που είμαι διοκτήτης αυτής της τηλεόρασης, τη τηλεοπτική αυτή συσκευή πηγαίνω στο δικαστήριο για να την προσβάλλω την απόφαση αυτή. Άρα, αν δεν υπάρχει απόφαση δικαστή, δεν μπορείτε να κατάσχετε, να δημεύσετε τίποτα. Καμία περιουσία. Κανένα περιουσιακό στοιχείο. Με απόλυτη ηρεμία μας λέει η Κομισιόν, α, δεν υπάρχει πρόβλημα εδώ. Επόμενο σημείο. Υποχρέωση του καταναλωτή να έχει δημόσια τηλεόραση και στη Ρουμανία. Και στην Ιταλία βέβαια ισχύει αυτό. Ακόμη και αν πληρώνουν για ένα συνδρομητικό ίσως ε, σταθμό, για άλλες υπηρεσίες, τουλάχιστον στη χώρα μου οι πολίτες έχουν πάρα πολύ, ε, πολλές δυνατότητες ε, για τη δορυφορική καλωδιακή τηλεόραση. Υπάρχει μεγάλη διείσδυση καλωδιακής τηλεόρασης. Αν λοιπόν εγώ θέλω να πάρω συνδρομή σε ένα τέτοιο ε, πάροχο, θα μου προσφέρει μεταξύ άλλων και κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης. Και θα έχω το μηνιαίο τιμολόγιο αυτού του ιδιωτικού παρόχου, υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης για τις υπηρεσίες που αγόρασα. Αλλά αυτό πρόκειται αυτό είναι ένα συμβόλαιο που έχω εγώ υπογράψει με αυτόν τον ιδιωτικό πάροχο. Που τον πάροχο δεν τον ενδιαφέρει αν εγώ ε, τη χρησιμοποιώ την υπηρεσία του ή όχι. Άμα πληρώνω, είναι ικανοποιημένο αφού έχουμε αυτή τη σύμβαση, αυτό το συμβόλαιο. Πώ λοιπόν είναι δυνατόν να αγοράζω εγώ αυτή τη δέσμη υπηρεσιών, αυτό μπουκέτο καναλιών από έναν ιδιωτικό πάροχο και μετά έρχεται δημόσια τηλεόραση και μου λέει όχι πρέπει να πληρώσετε εξτρά. Δεν με ενδιαφέρει τι έχετε εσείς, τι συμβόλαιο έχετε. Δηλαδή πληρώνω δύο φορές την ίδια υπηρεσία. Δεν το βρίσκει αυτό η Κομισιόν μονοπωλιακό ως ε, σύστημα. Και μην ξεχνάτε ότι είμαι και σοσιαλιστής. Δεν είμαι νεοφιλελεύθερος ούτε υπέρμαχος ε, του άναρχου καπιταλισμού που μας έφερε και σε αυτήν την κατάσταση. Αν λοιπόν επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε το ευρωπαϊκό νομικό σύστημα θα αρχίσει να έχει μεγάλα προβλήματα. Ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να πω ότι όντα αντιμέτωποι με αυτήν την πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλύσει τα προβλήματα, τα νομικά που σα προανέφερα. Αυτή η χαλαρή απάτη που μας δώσατε δεν μας ικανοποιεί καθόλου. Πρέπει να υπάρχει ένας κανονισμός που θα έχει ευρωπαϊκή διάσταση, διότι δεν νομίζω ότι μόνο στην Ιταλία συμβαίνουν τέτοιου καταχρήσεις. Και κλείνω απευθύνοντας έκκληση να παραμείνει ανοιχτή αναφορά και να περιμένουμε μία επιτέλους πια σοβαρή ε, και εύστοχη απάντηση από την Κομισιόν. Αλλιώς η κοινή γνώμη θα στραφεί κατά των δημοσιοτηλεοπτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη εν γέννη. Και αυτό θα είναι κακό για τους κοινωνικούς μας στόχους. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τουργκάιθ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Υπήρξαν άλλωστε αρκετοί συνάδελφοι που εξέφρασαν αναλυτικά τις απόψεις τους για το θέμα αυτό και με πολλέ από τι απόψει που άκουσα από του συναδέλφου συμφωνώ. Αυτό όμω που κυρίω θέλω να τονίσω, νομίζω μια Ιταλίδα συνάδελφο το είπε, ότι δηλαδή η Κομισιόν δεν έχει εκφραστεί ξεκάθαρα για διάφορα ζητήματα που θέτουν στην αναφορά τους οι αναφέροντες. Προσπαθεί να υπεκφύγει δηλαδή η Κομισιόν ή να ξεφύγει τέλος πάντων. Δεν θέλω να ε, επαναλάβω αυτά που είπαν οι συναδελφοί, αλλά θα σας κάνω δύο αποδείξει. Πρώτη, επειδή υπάρχει και θέμα ελεύθερου ανταγωνισμού, το διαπιστώσατε και εσείς φαντάζομαι κυρία Πρόεδρε, ακούγοντας την απάντηση της Κομισιόν και τα αιτήματα των αναφερόντων. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η Επιτροπή μας θα πρέπει να παραπέψει το θέμα στην Επιτροπή που είναι αρμόδια για τα ζητήματα του ελεύθερου ανταγωνισμού, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Να αναλύσει δηλαδή και αυτή η Επιτροπή με το δικό της, από τη δική της οπτική γωνία. Να μας δώσει τη δική της γνωμοδότηση για το θέμα αυτό. Δεύτερη υπόδειξη. Λέγοντας αυτό είναι λογικό ότι εννοώ βέβαια ότι θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να εξετάζουμε και να μελετούμε αυτό το θέμα. Σε καμία περίπτωση, κυρία Πρόεδρε, δεν μπορούμε να κλείσουμε μια αναφορά που έχει πιο πολλέ σκιέ παρά φωτεινά σημεία μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ευχαριστώ κύριε Τουργκάης. Ο κύριος Μποργέτσιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η εκπρόσωπος της ΡΑΗ μα είπε διάφορα πράγματα, τα οποία σίγουρα τα, είχαν προετοιμάσει οι διάφοροι υπάλληλοι τη νομική υπηρεσία της ΡΑΗ, οι οποίοι ε, γεμίζουν διάφορους θόκους, έχουμε διάφορους δικηγόρους, νομικούς, τεχνικούς κτλ. που σειραίουν εκεί πέρα στη ΡΑΗ και καταλαμβάνουν θέσεις. Ε, και πρόκειται για ένα εθνικό σκάνδαλο το οποίο θα πρέπει να ακουστεί χειρά και να καταγγελθεί στην, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί για να τους πληρώνουμε αυτούς τους ανθρώπους ε, γίνονται θυσίες, ε, αυτοί οι κύριοι και αυτές οι κυρίες ε, πληρώνονται με παχυδούς μισθούς, ενώ ε, διάφοροι ε, συνταξιούχοι πληρώνουν το, το τέλος. Υποτίθεται ότι έχουμε, πληρώνουμε πούμε, για δημόσια τηλεόραση. Και όμως, πού είναι εδώ η δημόσια τηλεόραση, εδώ συζητάμε ένα πολύ σημαντικό θέμα που ενδιαφέρουν τους ε, ε, πολίτες, ε, τους Ιταλούς πολίτες που πληρώνουν αυτόν τον ντροπιαστικό φόρο. Αλλά πού είναι η ΡΑΗ εδώ μέσα. Δεν υπάρχει για να ενημερώσει τους Ιταλούς πολίτες για αυτή τη συζήτηση που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να η παραπληροφόρηση. Δεν υπάρχει επαρκή ενημέρωση. Ο Ρουμάνος Ευρωβουλευτής είπε πολύ σωστά όλα όσα γίνονται στη Ρουμανία. Θα μπορούσαμε να τα λάβουμε υπόψη αυτά τα στοιχεία. Η περίπτωση της ΡΑΗ μου υπενθύμησε ε, τα όσα έλεγε ένας μεγάλος στοχαστής της δεκαετίας του 60 ε, για τις ε, μαφιόζικες δημοκρατίες. Η περίπτωση της ΡΑΗ ακριβώς αυτό δείχνει. Υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία αποσιωπεί, γίνονται διάφορα πράγματα μάλλον, τα οποία αποσιωπεί η ΡΑΗ. Ε, αυτό είναι μαφιός και δημοκρατία. Μέσω ε, χρηματοδοτήσεων, μέσω δικαστών που έχει στην τσέπη κτλ. Ε, ρωτήστε την, πρόταση, την πρόεδρο, κυρία πρόεδρε, κύριε εκπρόσωπο της Επιτροπής, Πόσος χρόνος δόθηκε από τη ΡΑΗ στο να ακουστούν οι σωστές παρατηρήσεις και τα νόμιμα δικαιώματα αυτών που πληρώνουν το τέλος ε, ΡΑΗ ε, σε εκπομπές κτλ. Πρέπει να ντρέπεστε. Ευχαριστώ κύριε Μποργέζιο. Σαλβίνη. Grazie Presidente. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μου κάνει κατάπτυξη, όχι μόνο η υπεράσπιση από πλευρά ΡΑΗ, η οποία υπερασπίζεται τι, τα προνόμια της. Ε, αλλά κυρίως με εκπλήσει η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η επιφανειακή στάση της αυτή. Μιλάμε για ένα όργανο που καταγγέλει τους πάντες, ελέγχει πώς ε, παράγεται το γάλα, πώς φτιάχνεται το το τυρί ας πούμε, πώς ψαρεύουμε ας πούμε στην, ε, στη Λιγούρια, καταγγέλει κάθε τρεις και λίγο ας πούμε τους πάντες και μπροστά σε αυτή την κατάφορη διάκριση που υφίστανται ε, οι χρήστες, ε, ειδικά όσοι έχουν αναπηρίες, τυφλοί, κουφοί κτλ. Ε, σε αυτά, σε αυτά τα, τα, προβλήματα κλείνει τα μάτια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλάμε για ανθρώπ, επίσης για άλλους ανθρώπους που πληρώνουν και που δεν, θα θέλανε να δεν μπορούν να λάβουν το σήμα της ε, ΡΑΕ. Θα ήθελα η Ευρώπη να καταψηφίσει, οι Ευρωπαίοι πολίτες να καταψηφίσουν αυτή την Ευρώπη. Υπάρχει μια τρύπα στη ΡΑΗ, δεκάδες ε, χιλιάδες ευρώ, Συχνά ε, βλέπουμε εκπομπές, εκπομπές οι οποίες θα μπορούσαν να τις κάνει και ο γιος μου που είναι 10 χρονών ας πούμε και παίρνουν εκατομμύρια ευρώ. Αγνοούν οποιαδήποτε ευρωπαϊκή δραστηριότητα. Οι, οι, συζητήσεις που κάνουμε εμείς εδώ και πώς εκπροσωπούνται στη ΡΑΗ, ποια είναι. Ο τρόπος εκπροσώπησης είναι, παρουσίασης μάλλον είναι απαράδεκτος. Για να μην πω δεν υπάρχει. Επίσης, οι τοπικές γλώσσες αγνοούνται, οι περιφερειακές απόψεις αγνοούνται. Υπάρχει μια απίστευτη έπαρση απέναντι σε αυτούς που δίνουν μάχη για να μην πληρώσουν αυτή την, αυτό το φόρο που είναι μια απάτη. Υπάρχουν ε, πολλά άλλα κανάλια που δίνουν αυτή την υπηρεσία πολύ καλύτερα και δωρεάν. Κανένα όμω δεν μπορεί να αγγίξει το ράιλ, όπω λέει η Επιτροπή. Όσοι δεν βλέπουν, πληρώνουν. Δεν έχουν όμω υπηρεσία. Οι κουφοί πληρώνουν και δεν έχουν υπηρεσία. Εκατομμύρια άνθρωποι πληρώνουν και δεν βλέπουν την. Ε, οι τυφλοί πληρώνουν και επίση δεν, ε, δεν βλέπουν τη ράιλ. Αλλά εσεί μα λέτε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τη ράιλ. Σας παρουσιάζουμε ένα τόνο έγγραφα και εσείς ούτε που δίνετε σημασία τα αγνοείται πάντελος και οι χιλιάδες υπάλληλοι της ΡΑΗ που κάνουν που υπάρχουν οι περισσότεροι υπάλληλοι της ΡΑΗ, μιλάμε για χιλιάδες άτομα, ε, κερδίζουν πολλά λεφτά και δεν κάνουν τίποτα. Υπάρχουν ελάχιστοι οι οποίοι πραγματικά κάνουν φοβερή δουλειά και θα πρέπει να πληρώνονται τριπλά, αλλά είναι λίγοι. Τέλο πάντων, καθένα έχει την τηλεόραση που του αξίζει. Ίσως η Ιταλία τη αξίζει να έχει μια τέτοια τηλεόραση. Θα ήθελα να ακούσω ε, απόψεις από άλλες χώρες, από άλλες κοινωνίες, από άλλους πολιτισμούς. Υπάρχει δημόσια τηλεόραση ε, ή δεν υπάρχει δημόσια τηλεόραση. Ε, εκτός και αν μας δουλεύετε. Μάλλον δεν είναι πολύ έξυπνη οι Ιταλοί μάλλον είναι λίγο βλάκε, αλλά και οι βλάκε ακόμα εξεγείρονται κάποια στιγμή. Ευχαριστώ κύριε Σαλβίνη. Δεν ζητάει κανένα άλλο το λόγο. Ζητάω καταρχήν, αν θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει στα ερωτήματα που ακούστηκαν, πολλά ερωτήματα, ειδικά ε, σε σχέση με τα νέα στοιχεία που παρουσίασαν οι εκπρόσωποι της Ιταλίας για το θέμα της ΡΑΗ. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι εκπλήσωμε από το ύφος κάποιων από τις παρεμβάσεις που άκουσα εδώ. Καταλαβαίνω πάντως απολύτως ότι υπάρχει θυμός από πλευράς πολιτών ε, για ε, ένα τέλος ε, που πρέπει να πληρώσουν για κάτι που δεν θέλουν να δουν ή που θεωρούν ότι είναι χαμηλής ποιότητας. Και πάλι όμως αυτό δεν είναι πρόβλημα που αφορά τις κρατικές ενισχύσεις. Αποτελεί εθνικό πρόβλημα. Το πώς καθορίζεται η χρηματοδότηση της δημόσιας τηλεόρασης. Καταλαβαίνω ότι στη Ρουμανία εφαρμόζεται διαφορετικό σύστημα. Ότι υπάρχει αμοιβαία συμφωνία, δηλαδή δηλώνει κανείς ότι εγώ θέλω να, πληρώνω, να, θέλω να βλέπω δημόσια τηλεόραση, άρα την πληρώνω. Ε, αυτό είναι άλλο μοντέλο. Τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να επιλέξουν ποιο μοντέλο θα εφαρμόσουν. Υπάρχει και ένα θέμα που τέθηκε σχετικά με κυρώσεις για όσους δεν θέλουν ή δεν μπορούν να πληρώσουν τα τέλη. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι σκληρές τέτοιες κυρώσεις, αλλά ξεφεύγουμε έτσι από το θέμα της δημόσιας τηλεόρασης και του σχετικού τέλους. Είναι κάτι που έχει να κάνει με κυρώσεις για πολίτες που δεν συμμορφώνονται με τους εθνικούς κανόνες. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού δεν θέλει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό, δεν νομίζω ότι έχουμε σχετική εντολή. Πρόκειται και πάλι για εθνικό θέμα. Επίσης, αναφέρθηκε απόφαση, πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ε, δεν την γνωρίζω. Εάν μου δώσετε αντίγραφο, πολύ ευχαρίστω θα την εξετάσω. Ευχαριστώ. Ακούσατε την απάντηση της Επιτροπής, που φαντάζομαι ότι δεν είναι επαρκή σε σχέση με τα ερωτήματα που ακούστηκαν. Αναγκαζόμαστε λοιπόν από πλευρά Προεδρία να υποβάλουμε γραπτό αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ακούστηκαν κάποια επιχειρήματα για κάποιες παραβιάσεις, τα οποία δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αναπάντητα, ξεκινώντας από την παραβίαση, την υποτιθέμενη παραβίαση, για την, α, τις διατάξεις της οδηγίας προστασίας του καταναλωτή. Ε, επίσης, ε, προβλήματα παραβιάσεων για την ε, ελευθερία του πολίτη όταν σφραγίζεται η τηλεοπτική συσκευή. Και επίσης, για δεδομένα τα οποία δεν έχουν καταλάβει σωστά από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μιλάμε για πολίτες που δεν θέλουν να βλέπουν τη ΡΑΗ, αλλά για πολίτες που είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη ΡΑΗ και να θέλαν. Όσο κακό και να είναι, όσο κακή και να είναι η ΡΑΗ και τα κανάλια και τα προγράμματα, και να θέλαν δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, να τα δούνε. Αυτό λέμε, δεν το κατάλαβαν μάλλον οι πρόσωποι τη Επιτροπή. Ο κ. Μποργέτσιο θέλει να πάρει το λόγο. Χωρί μικρόφωνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα έλεγα να προσθέσετε και κάτι άλλο στα όσα αναφέρατε. Μια πρόσκληση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαληθεύσει εάν υπάρχει προστασία επαρκής προστασία των γλωσσικών μειονοτήτων, όχι μόνο των διαφόρων περιφερειών, ειδικά της Βόρειας Ιταλίας που εκπροσωπεί το κίνημά μου, αλλά όλων των ε, Ιταλικών περιοχών. Ε, ξέρετε πολύ καλά ότι στη χώρα μας οι γλωσσικές μειονότητες είναι ένας απίστευτος πολιτιστικός ε, θησαυρός και μια απίστευτη παράδοση. Υπάρχει σοβαρότητη παραβίαση της υποχρέωσης που αναφέρεται και στις ευρωπαϊκές οδηγίες επαρκούς προστασίας για την προστασία, όχι μόνο πολιτιστική, αλλά του δικαιώματος έκφρασης ε, σε μία μειονοτική γλώσσα. Δικαίωμα το οποίο δεν προστατεύεται. Ευχαριστώ κύριε Μποργέτσιο. Ένα λεπτό θα δώσω στην κυρία Μαρτορέλη από πλευράς ΡΑΗ για να απαντήσει. Ευχαριστώ. Θέλω να σταθώ μια στιγμή, όχι σε όλα τα σημεία είναι αδύνατον, αλλά σε αυτό που υπόθηκε από, τον, από τους ευρωβουλευτές για την απόφαση του Αυγούστου του 2013 το Συμβούλιο Επικρατείας. Αυτό το σημείο προβλεπόταν στην ε, αναφορά. Στο... Όταν ε, έλεγε η σύμβαση της ΚΑΙ Ιτάλια, η ΡΑΙ ε, όλο το προγραμματισμό της δημόσιας τηλεόρασης, όλα τα προγράμματα, τα έβαλε σε μια πλατφόρμα τη που δημιουργήθηκε το 2009 και τέθησε στη διάθεση των ε, χρηστών. Είναι μια πλατφόρμα δορυφορική. Μην ξεχνάτε ότι η χερσαία ψηφιακή τηλεόραση, που είναι η βασική τηλεόραση, ε, καλύπτει τα 4 πέμπτα του πληθυσμού. Και μόνο ένα πέμπτο του πληθυσμού ε, έχει δορυφορική λήψη. Η ΡΑΗ δεν υποχρέωσε με αυτόν τον τρόπο ε, τους χρήστες της να πληρώσουν μέσω συνδρομής την υπηρεσία αυτή Sky. Επομένως η TV SAT λαμβάνεται από τους χρήστες μέσω ε, μια συσκευή setup box. Η Sky ε, έκανε αυτή την, έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Και με βάση την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας του 2013 δεν υπάρχει υποχρέωση από την ΡΑΗ να δώσει δωρεάν τα προγράμματα, του, τα προγράμματα δημόσιας τηλεόρασης. Και στο τέταρτο εδάφιο του άρθρου 22 ε, της σύμβασης της ΡΑΗ προβλέπεται η δυνατότητα από τη ΡΑΗ να δώσει ε, σε διάφορους εμπορικούς φορείς ε, τη δυνατότητα να, να αναμεταδίδει τα προγράμματα με βάση ε, συγκεκριμένους όρους, μη, χωρίς διακρίσεις και τέτοια. Ε, επομένως τα προγράμματα αυτά θα μπορούσαν να Αυτά τα προγράμματα που δίδονται στο Sky ε, δίδονται με ένα κωδικοποιητή. Η, πλατφόρμα αυτή που έδωσε, στη, ε, που η ΡΑΗ, η TVSAT, συνάδει με μια αντίληψη ε, δυναμική, εξελικτική της δημόσιας τηλεόρασης. Και δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα ε, σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις και με, τις, με την παροχή υπηρεσιών κοινή ωφελίας. Όλα τα υπόλοιπα δεν πρόλαβα να τα πω. Ένα λεπτό για την απάντηση δίνω στους εκπροσώπους των συνταχτών της αναφοράς. Θα μιλήσω εγώ και θα τους εκπροσωπήσω όλους τους συντάκτες. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είδε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η ΡΑΗ την είδε, αλλά την ερμηνεύει λάθος. Η Sky είχε προσφέρει 350 ε, εκατομμύρια ευρώ στη ΡΑΗ, το υπενθυμίζω, για να μπορεί να, να μεταδίδει τα προγράμματα ΡΑΗ. Αυτό το ξέρει η εκπρόσωπος της ΡΑΗ, είμαι σίγουρη. Σας παρακαλώ διαβάσετε καλά την απόφαση του ελεγκτικού του Συμβουλίου της... Ε, e το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και ζητάω από την πρόεδρο Ματσόνη, μια και είναι έτσι κατάσταση, αν μπορείτε, και μια και γίνεται μια τρομερή συζήτηση στην Ιταλία, αν μπορείτε να έχετε σε επαφή με την Επιτροπή Εποπτείας της ΡΑΗ, για να καταλάβετε για ποιο λόγο ο πρόεδρος έκανε κατάληψη και εξακολουθεί να κάνει κατάληψη στη ΡΑΗ αυτή τη στιγμή, ο διευθυντής μάλλον. Μιλάμε τώρα για το φορέα ο οποίος αποπτεύει και ο οποίος κάνει κατάληψη στην, στη ΡΑΗ. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ασχοληθεί με το δικαίωμα ενημέρωσης όλων των πολιτών. Νομίζω ότι είναι καλό αυτό, καθάστε να ενημερωθείτε εσείς και να ενημερωθούν και όλα τα υπόλοιπα ε, κράτη εν συνεχεία. Ευχαριστώ. Να συνοψίσω τη συζήτηση, όπως την αντιλαμβάνει η Προεδρία, εμείς ως Επιτροπή Αναφορών έχουμε το δικαίω... την υποχρέωση να ακούσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες και να δώσουμε απαντήσεις στα αιτήματά τους. Σε σχέση με αυτή την αναφορά που μόλις εξετάσαμε, έχουμε το καθήκον να προχωρήσουμε εις βάθος για να καταλάβουμε αν πραγματικά υπάρχει παραβίαση, όπως κατήγγειλαν οι συντάκτες της αναφοράς, και αν όλα αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούσαμε σήμερα στην αίθουσα ε, έχουν βάση. Επομένως, έχω το, την υποχρέωση να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχω το, το δικαίωμα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξαναδεί αυτό το θέμα για να δει αν υπάρχει κάποια παραβίαση εδώ. να εξετάσει ενδεχομένως όλα τα θέματα και να δει πώς μπορεί να προστατεύσει τους Ευρωπαίους πολίτες. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας, αυτός ο οποίος κάνει κατάληψη στα κτίρια της ΡΑΗ, εξέφρασε κάποια προβλήματα, κάποια επιχειρήματα. Ίσως καλό θα ήταν να έρθουμε σε επαφή με την Επιτροπή αυτή εποπτείας για να καταλάβουμε ποια είναι τα όρια ανάμεσα στα όσα μπορούμε εμείς να προστατεύσουμε και στα όσα εποπτεύει αυτή η Επιτροπή Εποπτείας. Ζητάω λοιπόν τους συναδέλφους να μην κλείσει αυτή η αναφορά, ούτω ώστε να μπορέσουν να δώσουν μια απάντηση. Πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί απάντηση. Δεν έχει δοθεί με τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ούτε μετά όσα μας είπε η εκπρόσωπος της ΡΑΗ είμαστε ικανοποιημένοι. Ας κρατήσουμε λοιπόν ανοιχτή αυτή την αναφορά. Δεν ξέρω αν συνόψα καλά τη συζήτηση. Ε, σας ρωτάω, συμφωνείτε με αυτή την πρόταση. Δεν βλέπω αντιρρήσεις. Επομένως, συμφωνούμε με την πρόταση να συνεχίσει η αναφορά όπως ε, ακούσατε από μένα. Ευχαριστώ τους συντάχτες, ευχαριστώ την υπεύθυνη της ΡΑΗ για την παρουσίασή της και περνάω στην επόμενη αναφορά. Η επόμενη αναφορά ποια είναι. Είναι το, αυτή στο σημείο 7. Συν Λόλες, Ιρλανδός πολίτης, αφορά μια αναφορά σχετικά με ασφαλμένη εφαρμογή των όρων και προποθέσεων για τα συστήματα ενιαία ενίσχυσης, αναγεωργική εκμετάλλευση και μειονεκτική περιοχή στι αρχέ του Galway στην Ιρλανδία. Η κυρία Μέρφυ θα πάρει το λόγο που εκπροσωπεί του συντάκτες. Πρόεδρε, η αναφορά αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της ε, του ότι ε, οι Ιρλανδικές ε, αρχές ε, δεν εφαρμόζουν σωστά το σύστημα ενιαίας ενίσχυσης αναγκαιορική εκμετάλλευση και μειονεκτική περιοχή. Η εν λόγω έκταση βρίσκεται σε μια ειδική προστατευμένη περιοχή για πουλιά και η οι εκτάσεις αυτές είναι παρόμοιες με τις γειτονικές και οι επιθεωρητές ε, έχουν παραστεί σε διάφορες επιθεωρήσεις ε, οι οποίες όμως ε, δεν έχουν ανακοινωθεί στους μετόχους. Έχει καθοριστεί η κτηνοτροφική αναφορά 95% η οποία μειώθηκε στο 0% και μετά αυξήθηκε στο 10%. Άλλες γειτονικέ εκμεταλλεύσεις με παρόμοια χλωρίδα έχουν επιθεωρηθεί επίσης και ε, έλαβαν κοινοτροφική αναφορά άνω το 95%. Και οι μέτοχοι ε, ανησυχούν για τη διακριτική αυτή μεταχείριση. Ε, θέλουμε λοιπόν το, για τα έτη 2010 Κάποιοι μέτοχοι έχουν λάβει πλήρη πληρωμή για το 2010, 2011 και 2012, ενώ ε, άλλοι καθόλου. Επίσης, ε, ένας από αυτούς ε, ζήτησε να μάθει γιατί δεν, δεν έχει γίνει η καταβολή των χρημάτων. αλλά του είπαν ότι δεν... Παρακαλώ κυρία Μέρφη, πιο αργά λέει η πρόεδρος. Ο μέτοχος ε, πληρώθηκε χωρίς ε, καμία εξήγηση μετά από τα παραπονά του, μια διαδικασία με την οποία θα έχανε σημαντικές πληρωμές ε, στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών υπό το φως της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής και της μεταρρύθμισής της. Άλλος μέτοχος Ε, προς τον οποίο ανακοινώθηκε η κοινοτροφική αναφορά ε, ύψους 10% ζήτησε να προσφύγει κατά της ε, διαδικασίας αυτής με βάση την, διαδικασία, την εσωτερική διαδικασία προσφυγής η οποία ξεκίνησε το 2010 και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο ετών δεν μπορεί να λάβει αποζημίωση διότι δεν μπορεί να χειριστούν τα δικαστήρια τα θέματα, το θέμα αυτό προτού να ε, ολοκληρωθεί η διαδικασία προσφυγής. Υπολογίζεται ότι μπορεί τρία χρόνια να απαιτηθούν για να φτάσει η διαδικασία σε αυτό το στάδιο και αυτό είναι κάτι που επηρεάζει όλους τους μετόχους ε, με παρόμοιο τρόπο. Όσο περνάει ο χρόνος, ε, το Υπουργείο αυξάνει την οικονομική πίεση. Γιατί λοιπόν ζητάμε να παρέμβει η Επιτροπή Αναφορών. Γιατί δεν μπορεί να ε, ε, ε, ασκηθεί δικαστική δίωξη στο κράτος μέλος. Η διαδικασία εντό των κρατών μελών μπορεί να απαιτήσει πάνω από πέντε χρόνια, κάτι που σημαίνει ότι με την έναρξη της διαδικασίας αποκλείεται ο ετών να ξεκινήσει η δικαστική προσφυγή. Και η υπερβολική καθυστέρηση καθιστά αναποτελεσματική τη διαδικασία και έτσι ε, δεν μπορεί να βρει το δίκαιο του ο ετών. Υπό τις ε, συνθήκες αυτές απομένει μόνο η δυνατότητα να αγνοηθεί η διαδικασία προσφυγής και να ξεκινήσει η δικαστική προσφυγή. Γιατί ζητάμε την παρέμβαση της Επιτροπής Αναφορών. Ο κ. Μάικ Μέρφυ, στον οποίο αναφέρθηκα και πιο πριν, που είναι μέτοχος, ε, ξεκίνησε διαδικασία προσφυγής, η οποία όμως αγνοήθηκε τελείως ε, από τη σχετική αρχή. όπως επίσης ε, δεν του δόθηκαν εξηγήσεις ε, γιατί ε, μειώθηκε η κτηνοτροφική αναφορά στο 10%. Έπρεπε να έχει πληρωθεί για το 2010 και 2011, 2012 και 2013 τώρα. Η αρχή ε, ζήτησε να λυθεί το θέμα πληρώνοντας τον, ε, ε, τα χρέη με βάση μια επανεξέταση που έγινε τον Ιανουάριο του 2013. Μέσω του δικηγόρου συμφώνησε να αποσύρει την προσφυγή εφόσον πληρωθούν και τα νομικά έξοδα. Ενημερώθηκε γραπτός από ε, την ε, αρχή ότι μπορεί να προσφύγει ε, κατά της ενοποίησης των δικαιωμάτων που είχε. Μέχρι στιγμής δεν έχει εξεταστεί η προσφυγή του. Όχι μόνο είναι απίστευτα κακή πρακτική αυτή, αλλά είναι ενδεικτική και της στάσης της ε, αρμόδιας αρχής απέναντι στους ε, αγρότες που ε, που προσέφηκαν στα Ιρλανδικά δικαστήρια. Ξέρω ότι η αρχή της Επιτροπής σας είναι ότι αυτή η υπόθεση θα πρέπει να εξεταστεί από τα Ιρλανδικά δικαστήρια. Αλλά ε, νομίζω ότι σας έχω δείξει ότι ε, η αρμόδια αρχή έχει μπλοκάρει τις διαδικασίες ε, και εσωτερικής προσφυγής και δικαστικής προσφυγής. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βρίσκονται ανάμεσα στη σκύλα και στη χάριβδη οι αγρότες και Η θέση τους έχει ε, καταστεί ιδιαίτερα δυσμενής. Ε, τι ζητάμε λοιπόν από την Επιτροπή Αναφορών να κάνει για μας. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ε, οι μέτοχοι ανα πάσα στιγμή δέχτηκαν το προνόμιο της Δημόσιας Αρχής να μειώσει την επιλεξιμότητα των εν λόγω εκτάσεων εφόσον αυτό συνάδει με την αντιμετώπιση παρομοίων εκτάσεων στην Ιρλανδία και σε όλη την Ευρώπη. Σε, γι' αυτό το λόγο σας ζητάμε ε, να εξετάσετε την ε, υπόθεση και θέλουμε δίκαιη ε, αντιμετώπιση και μια ανεξάρτητη έρευνα. Θέλουμε η γη να εξεταστεί ως προς την επιλεξιμότητά της από επιθεωρητή τελείως ανεξάρτητο από το Υπουργείο ε, Γεωργίας της Ιρλανδίας. Ε, δράσεις που αναλαμβάνουν τα ε, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είχαν τεράστιο αντίκτυπο όσον αφορά την δίκαιη εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. Ζητάμε από την Επιτροπή Αναφορών ε, να ε, συνεχίσει την, ε, την αφοσίωση της στα θέματα αυτά, να υπάρχει έτσι δικαιοσύνη και αμεροληψία, σωστές διαδικασίες σε περιπτώσεις προσφυγής που αφορούν τέτοιες εκτάσεις. Επίσης, ζητάμε οι υπάλληλοι του Υπουργείου να πρέπει να λογοδοτήσουν για την, ε, για την μη σωστή εφαρμογή του προγράμματος αυτού. Πολύ ευχαρίστω θα απαντήσω σε ερωτήσεις. Thank you. now the floor... Σας ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Βαλεριάτου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως ακούσατε, η αναφορά αφορά την εφαρμογή ενιών πληρωμών ή ενισχύσεων ε, μειονεκτικών ε, περιοχών από ένα κράτο μέλο δυνάμει τη κοινή γεωργική πολιτική. Ακούσαμε από την αναφέρουσα ένα πρόγραμμα εφαρμογής ε, και αξιολόγησης των επιλέξιμων για αυτή την ενίσχυση εκτάσεων από ένα κράτος μέλος. Μιλάμε λοιπόν για την εφαρμογή αυτών του καθεστώτος ενός πληρωμών και αυτό είναι ευθύνη των κρατών μελών, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Το έχουμε πει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αξιολόγηση ε, της αναφοράς, ε, της επιλεξιμότητας ε, των γεών είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών που υποτίθεται πρέπει να εφαρμόζουν την κοινή γεωργική πολιτική. Δεν μπορεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποκαταστήσει την αξιολόγηση της κατάστασης δεν μπορεί να υποκαταστήσει αυτή την αξιολόγηση των επιλέξιμων εκτάσεων και των χορτονομών. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί στη διαφορά αυτή ε, μία λύση ενώπιον όμως ε, των εθνικών ε, διοικητικών αρχών. Η αναφορά αφορά, να αναφέρει επίσης και την δυνατότητα ή μη δυνατότητα δικής δίκης, αλλά και αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών της ευθύνης της εθνικής, άρα η λύση θα πρέπει να αναζητηθεί ενώπιον των εθνικών αρμόδιων αρχών. Παραμένω στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χίγγινς έχει το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα καλωσορίζω τους συναδέλφους από την Ιρλανδία. Η κυρία Μέρφη νομίζω τα είπε πάρα πολύ πιστικά σε ό,τι αφορά αυτά που συμβαίνουν εδώ στην προκειμένη περίπτωση. Θέλω να ξανασυνοψίσω. Δεν υπάρχει δυνατότητα έφεσης. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Άρα φανταστείτε ότι απαιτούνται πέντε χρόνια για μια έφεση τι θα κάνει στο ενδιάμεσο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος. Πώς θα ε, αποζημιωθούν. Είναι τρελές αυτές οι προθεσμίες. Πώς έχει κατάσταση κύριε Πρόεδρε. Εν λόγω κτηνοτρόφοι λάμβαναν 99% των πληρωμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και γίνονταν ετήσια ε, έλεγχοι. Από τη μια μέρα στην άλλη όμως ε, έτσι γιατί το αποφάσισε το Υπουργείο Γεωργίας, αναστάλησαν οι πληρωμές. Και όταν υπήρξαν εφέσεις, οι προσφυγές, ε, η πληρωμή ε, που επαναλήφθηκε ανερχόταν σε 10% μόνο. Είναι τρελό κάτι τέτοιο. Πρέπει οι ενισχύσεις να δίνονται ξεκάθαρα στους ε, κτηνοτρόφους με σαφές κατευθυντήριες γραμμές που ναι μεν παλιά ήταν, ε, ε, μετά επειδή υπήρξε αυτή η απόσταση των ενισχύσεων και η νέα ε, καταβολή του σε πολύ μικρό τρόπο σωστό υπάρχει κακή διαχείριση. Και πολλές φορές οι πληρωμές αυτές έχουν ταπανηθεί πολύ πριν ληφθούν, επειδή γίνεται μια πρώιμη απελευθέρωση αυτών των ποσών από την Ιρλανδία. Πρέπει λοιπόν να γίνουν διάφορα πράγματα. Πρώτα απ' όλα θέλω η Επιτροπή Αναφορών, που είναι πολύ αποτελεσματική στη δουλειά της, να γράψει στο Υπουργείο Γεωργίας ε, που ο Υπουργός του τυχαίνει να είναι και πρώην μέλλον σε της ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να πούμε ότι ε, δεν θεωρούμε ότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο να γίνεται η διαχείριση της γεωργικής πολιτικής γιατί μιλάμε για τις ζωές και την επιβίωση των γεωργών και των κτηνοτρόφων. Επίσης πρέπει να αναθέσουμε μια ανεξάρτητη επιροθεώρηση έλεγχο, όπως έκανε και η κυρία Μέρφη, ε, για να δούμε ακριβώς αυτή την κοινή χρήση των χορτοτόπων, των ε, χορτολιβαδιών. Διότι είναι τρομερό να περιμένει κανείς πέντε χρόνια αν έχει προσφύγει, αν έχει εφεσιβάλει την απόφαση. Υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές. Θέλω λοιπόν να ζητήσω από ε, το Υπουργείο να αναθεωρήσει αυτή τη ε, διάταξη. Τέλος, καλό, κυρία Πρόεδρε, την Επιτροπή μας να έρθει στην οπότε οποτεδήποτε και η Πρόεδρος ε, η Γραμματεία, να έρθετε λοιπόν στην Ιρλανδία όποια εποχή του χρόνου για να επισκεφτείτε αυτή την ε, έκταση, το Kildare, που το έχω επισκεφτεί προσωπικά και έχω δει την κατάσταση και μπορώ να σας πω ότι ακριβώς το διπλανό λιβάδι παίρνει αυτή την αποζημίωση του 90%. Εδώ βλέπετε αυτό τον χορτότοπο, αυτό το χάρτη. Και δίπλα βλέπουμε κάποιες ε, επιθεωρημένες εκτάσεις που παίρνουν εκεί το 90% της επιδότησης. Ε, αλλά αυτούς τους, ε, ε, τους τις πήραν πίσω όλες τις πληρωμές. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν κύριε Πρόεδρε που δεχθήκατε την αναφορά ε, Νόλης Μέρφη. Και το δεύτερο που θέλω να ζητήσω είναι να έρθετε στην Ραδία ή τέλο πάντων να παρακολουθήσετε εκ του σε αυτήν την κατάσταση. Mrs. McInnes. You asked first. Κύριε Μαγκίνε, όποιος ζήτησε πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ καλωσορίζω τους συντάκτες δεν θα ήταν εδώ σήμερα αν δεν είχαν σοβαρό πρόβλημα, αλλά έχουν. Και εμείς ως εκπρόσωποι του λαού έχουμε την υποχρέωση να τους υποστηρίξουμε απλώς, αλλά να τους υποστηρίξουμε και επειδή έχουν επιχειρήματα σε αυτά που λένε. Ε, οι επίσημες αρχές δεν μπορούν να πάρουν αυτή την απόφαση. Το θέμα ε, είναι αρκετά υποκειμενικό, αλλά αυτή το παρουσίασαμε με αρκετή αντικειμενικότητα και είναι πολύ λογικό να απαντήσουμε στην, στα αιτήματα της κυρίας Μέρφυ ότι πρέπει να γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα για την επιλεξιμότητα αυτών των εκτάσεων. Είναι το ελάχιστο που, μπορούμε που πρέπει να κάνουμε. Επίσης, ε, συμφωνώ με τον ε, Jim Higgins σε ό,τι αφορά τη διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ μακροσκελής, πολύ αργή. Ε, οι άνθρωποι αυτοί εξαρτώνται από αυτήν την ιστορία και Υπάρχει διακριτική μεταχείριση εναντίον τους. Κάνω έκκληση στα μέλη της Επιτροπής Αναφορών να υποστηρίξουν την απόλυτα λογική πρόταση που έγινε από τους συντάκτες. Πιστεύω ότι αυτά που ακούσατε είναι αρκετά για να καταλάβετε την υπόθεση, αλλά αν δεν αρκούν αυτά, ε, επισκεφτείτε την περιοχή. μπορείτε να αποφασίσετε να πάτε στο Δουβλίνο, ας πούμε, τις επόμενες εβδομάδες. Κυρία Μαγκίνες, ευχαριστώ τους συντάκτες, δεν είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής, ήμουν στο παρελθόν. Έχω κάποιες παρατηρήσεις να κάνω για το τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, ενδιαφέρομαι για αυτό το θέμα, γιατί ε, έχω ασχοληθεί με την πρώην γεωργική ε, πολιτική και υπάρχουν φυσικά επιπτώσεις για το μέλλον των συντακτών, αλλά και γιατί με ενδιαφέρουν κιόλας επειδή είναι Ιρλανδοί. Υπάρχουν γύρω ε, θετικά θέματα, ε, κάποια συγκεκριμένα θέματα, αλλά και κάποια γενικά γύρω από την αναφορά. Υπάρχει ένας χάρτης δικαιωμάτων αγροτών. Δηλαδή, αντιμετωπίζονται με ειδικό τρόπο οι γεωργοί. Χρήσιμο θα ήταν ως Επιτροπή εμείς να δούμε αν έγινε σεβαστή ο χάρτη αυτό απέναντι σε αυτό το συντάκτη. Δεν νομίζω ότι έγινε. Θα ήταν χρήσιμο να το δούμε αυτό. Ε, με τι ανησυχίε που είπαν κι άλλοι ότι ένα σύστημα προσφυγών που χρειάζεται πέντε χρόνια για να αποφασίσει μερικέ φορέ είναι εντελώ απαράδεκτο. Θα πρέπει να έχουμε ένα καλύτερο σύστημα προσφυγών, ένδικων μέσων, εν πάση με πιο μικρέ προθεσμίε. Αυτό είναι ένα γενικό ε, σχόλιο που επηρεάζει όλου ούτω ή άλλω του γεωργού. Ε, και είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Σε σχέση τώρα με το συγκεκριμένο θέμα που μας απασχολεί, μπορώ να υποστρίξω την ιδέα να γίνει μια χωριστή και ειδική έρευνα, αλλά από την εμπειρία που έχω από την Επιτροπή Αναφορών, όπου δίδουμε υποσχέσεις στους συντάκτες αλλά δεν τις στηρούμε, η εμπειρία μου δεν είναι θετική. Να μην δίνουμε υπερβολική έμφαση στο τι μπορεί να πετύχουμε εδώ, γιατί δεν έχουμε και αρμοδιότητες σε αυτόν τον τομέα ούτως ή άλλως. Να μην δίνουμε έμφαση λοιπόν σε αυτόν. Ίσως είναι πέραν της εντολής μας ε, το να διενεργήσουμε μια ανεξάρτητη έρευνα, παρότι χρειάζεται στην πραγματικότητα. Επομένως πρέπει να δούμε πώς η Κομισιόν μπορεί να βοηθήσει, η Επιτροπή μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το θέμα και όταν το κράτο μέλο είναι αρμόδιο σε αυτό το τομέα, όπως είπε και η Επιτροπή, ε, μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο το ελεγκτικό συνέδριο. Μπορεί να τσεκάρει και να ελέγξει αν εφαρμόζεται σωστά το σύστημα στον λόγο κράτο μέλο. Και αν, όταν υπάρχουν ερωτηματικά, όπως σε αυτήν την περίπτωση, κάποιο να τα κοιτάξει τουλάχιστον. Να μην είναι ο ίδιο δικαστή και δικαζόμενο, α πούμε, όπως ε, σε αυτήν την περίπτωση είναι το Υπουργείο Γεωργίας. Ας δούμε λοιπόν ποιος μπορεί να κάνει αυτή την ανεξάρτητη έρευνα, να βάλουμε κάποια χρονικά περιθώρια, κάποια προθεσμία, γιατί φοβάμαι ότι θα γίνει και εδώ όπως με προηγούμενες αναφορές. Δηλαδή είχαμε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που πέρασε από τη στιγμή που ξεκίνησε η υπόθεση μέχρι το συμπέρασμα, που στην πραγματικότητα προκαλεί αυτό απογοήτευση παρά βοηθάει. Και ούτω ή άλλω αυτοί οι συντάκτε προσπάθησαν επιμακρών να λύσουν το πρόβλημα αυτό στην Ιρλανδία. Α προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε την ιστορία αυτή. Μία επιστολή, ίσω, όπω είπε και ο κύριο Τζιμ Higgins, είναι ο καλύτερο τρόπο να προχωρήσουμε για να δούμε ποια είναι τα στοιχεία, ε, να ασχοληθεί, να επιληθεί το αρμόδιο Υπουργείο. Και αυτό είναι πρώτο βήμα, ένα πρώτο βήμα. Θα μπορούσαμε λοιπόν η Κομισιόν να εξετάσει το κατά πόσο μπορεί να γίνει μια ανεξάρτητη έρευνα και αν μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο το ελεγκτικό συνέδριο. Αν δηλαδή πρέπει να ενημερωθεί για αυτές τις διαφορές, ε, για το πώς εφαρμόζονται τα ευρωπαϊκά, ευρωπαϊκοί μηχανισμοί και το γεγονός ότι δεν πληρώνονται χρήματα στους, στους αναφέροντες. Ε, δεν τους δόθηκαν λεφτά τα οποία πιστεύουν ότι δικαιούνται και αυτό συμβαίνει για μεγάλο χρονικό διάστημα τώρα. Ευχαριστώ κύριε Σχεγγίνς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος να σας ευχαριστήσω θερμά όπως και την γραμματεία που δεχτήκατε αυτή ε, την αναφορά. Ε, περιμένουμε να δούμε τι συστάσεις που μπορείτε να κάνετε. Πρέπει να πω ότι με απογοητεύει πολύ η απάντηση της Κομισιόν, ε, αλλά βέβαια είναι προβλέψιμη. η επικουρικότητα μερικές φορές τους βολεύει. όταν μιλάνε για πολιτική αερομεταφορών, ε, πολύ σε είπα τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Ε, μιλάμε για Ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκό χρήμα και η Κομισιόν ε, έχει λόγο όσον αφορά το πώς δαπανάτε το ευρωπαϊκό χρήμα. Ευρωπαϊκό χρήμα που προορίζεται για ανθρώπους που δυσκολεύονται να επιβιώσουν μπλοκάρονται από υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας και πιστεύω ότι ενδιαφέρει την Κομισιόν το συγκεκριμένο θέμα. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα τη Επιτροπής Αναφορών, ε, δεν θέλω να διαφωνήσω με τον συνάδελφο, αλλά ε, σε... έχω δει πολλά θετικά αποτελέσματα ε, εδώ στην Επιτροπή Αναφορών. Εγώ και ο συνάδελφός μου που επίσης είναι υπεύθυνο για την ε, σημερινή αναφορά. Ε, είχαμε υποβάλει ε, αναφορά σχετικά με τις, με τις δαπάνες περιαγωγών. Επίσης είχαμε θετικό αποτέλεσμα πριν κάποια χρόνια. όπου η Επιτροπή Αναφορών υπέβαλε συστάσεις προς την Ιρλανδική κυβέρνηση. Η Επιτροπή, σας, ε, η Επιτροπή Αναφορών λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που δεχτήκατε αυτές τις αναφορές ε, και προσλέπουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ζητάει κανείς άλλο το λόγο. Η κυρία Μαγκίνε, ένα λεπτό, όχι παραπάνω. 30 δευτερόλεπτα, κυρία Πρόεδρε. Ο Τζιμ έχει δίκιο. Ε, ε, είδαμε σημαντική επιτυχία σε κάποιε αναφορέ. Είχαμε όμω και μια άλλη ε, αναφορά γεωργία, Νταν Μπρέναν, και νιώθω ότι παρότι σημειώνουμε κάποια πρόοδο, ο αναφέρον σε έχει περάσει από μακρά διαδικασία και καταβάλαμε προσπάθειες. Δεν νομίζω ότι δεν προσπαθήσαμε, αλλά δεν καταφέραμε πολλά. Εάν λοιπόν θέλουμε να βοηθήσουμε και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να θέσουμε ε, χρονικά όρια. Δεν αποτελεί επίκριση αυτό, γεγονός αποτελεί. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ, ναι, πράγματι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δέκα δευτερόλεπτα. διάβασα το θέμα αυτό και όποιες και να είναι οι νομικές δεσμεύσεις υπάρχουν ηθικές δεσμεύσεις ε, καθώς και ε, συμβατικές διότι οι άνθρωποι αυτοί ε, μπορεί να έχουν επενδύσει με βάση ενός εγγυημένου εισοδήματος το μνημόνιο κατανόησης υπάρχει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας αφιερώσατε το χρόνο σας. Ευχαριστώ. Ωραία. Δίνω το λόγο στην κυρία Μέρφη για ένα λεπτό για να απαντήσει. Νομίζω ότι ε, οι κύριοι Χέικινς, Μακάρι και Κάλαχαν ε, ε, έθιξαν όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν το, τους αναφέροντες. Είναι ένα θέμα όπου έχουμε συναντήσει εμπόδια σε κάθε κατεύθυνση και γι' αυτό αναγκαστήκαμε να προσφύγουμε στην Επιτροπή σας. Αυτό μόνο έχουμε να προσθέσουμε αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, ομόφωνο αίτημα να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή και να ε, στείλουμε επιστολή στον ε, Ιρλανδό Υπουργό Γεωργίας για να γίνει έρευνα. Μάλιστα μπορούμε να παραπέμψουμε το θέμα και στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και στο τέλος, ε, όταν θα λάβουμε απαντήσεις ε, στα αιτήματά μας, μπορούμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά ακόμα και νέα θέματα, ε, νέες πτυχές. Συμφωνείτε με την πρότασή μου. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους αναφέροντες, ευχαριστώ όλους για την ενδιαφέρουσα αυτή συζήτηση. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. που είναι η αναφορά 760 του 2007, σημείο 9 στην Μερσιά Διάταξη, από τον Κόζιμο Φρακάσο Ιταλικής Ταγένειας Και άλλους βέβαια. Πρόκειται για προειδοποίηση για διοξίνε στην πόλη Ταραντό. υπήρξαν νέα στοιχεία. Εξού και οι συνάδελφοι όπως η κυρία Άουκεν ζήτησαν να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή για να ξανακούσουμε τους εκπροσώπους των Ιταλών πολιτών. Σας υπενθυμίζω ότι για την εν λόγω αναφορά η Επιτροπή ξεκίνησε επιτέλους το Σεπτέμβριο, επιτέλους δικασία επιβολής κυρώσεων κατά της Ιταλίας. Δίνω το λόγο λοιπόν στην εκπρόσωπο. Θα μιλήσω αγγλικά, κυρία Πρόεδρε. Είμαστε εδώ μια σημαντική μέρα που αυτό το τρομερό θέμα της ε, μόλυνσης από διοξίνη είναι στο επίπεδο της προσοχή του Κοινοβουλίου, άρα και της κοινή γνώμη των Ευρωπαίων πολιτών. Το 2007 είχαμε υποβάλει αυτή την αναφορά για τις ε, διοξίνες. Ε, η πόλη της Ιταλία Ιταλίας, Τάραντο, από την οποία κατάγομαι και για την οποία βρίσκομαι εδώ, έχουμε δυστυχώς πολλές φορές ε, υποστεί ε, τα προβλήματα της διοξίνης. Είδαμε υψηλές συγκεντρώσεις της διοξίνης ε, πέρυσι, ίσως τις υψηλότερες στην Ευρώπη, αλλά στην πόλη μας πραγματικά δεν μπορεί να πει κανείς ότι ούτε τα ζώα ούτε οι άνθρωποι είναι στο απειρόβλητο. Και πολύ σύντομα ε, δεν θα μείνει τίποτα, γιατί κανένας δεν μπορεί να διατηρήσει την υγεία του, ούτε άνθρωπος ούτε ζώο, όταν έχουμε τέτοιου είδους υψηλές συγκεντρώσεις. Ε, η εταιρεία Ήλβα είχε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2013 στο επίκεντρο της προσοχής της κοινής γνώμης όταν κινήθηκε διαδικασία πολύ καιρός κατά της Ιταλίας που παραβιάζει την οδηγία για τις εκπομπές και για το ότι δεν σέβεται την περιβαλλοντική και για τη μη, μη των περιβαλλοντικών διατάξεων από την Ήλβα. Ο Γιάννης Ποτότσνικ, ο επίτροπο με πάρα πολύ γενναία επαγγελματική δράση, έδειξε, ε, έριξε τους διεθνούς, προβολή τη δημοσιότητα στην περίπτωση αυτή. Και έτσι το τάνατο έχει γίνει μια ευρωπαϊκή πόλη, ε, θέλουμε την υποστήριξή σας. Βρήκαμε ε, δύο ε, και στο μητρικό γάλα ακόμη, αλλά και ε, στον οργανισμό των ανθρώπων. 2.000 ε, ζώων ε, χρειάστηκαν ε, να σφαγούν λόγω της παρουσίας διοξίνης στα γαλακτοκομικά πρώτα και στο γάλα. Έγινε, διατάχθηκε έρευνα και βρέθηκε ομοιότητα μεταξύ του χημικού αποτύματος της διοξίνης στη Σίλβα με ένα αποτύπωμα στις περιοχές γύρω εκεί. Οι βοσκότοποι είναι πλέον απαγορευμένοι να χρησιμοποιούνται τα 10, στα, στη διάμετρο 10 χιλιόμετρων. Ε, αυτή η διοξίνη ε, ξέρουμε ότι παραμένει για πάντα και μολύνει ε, σιγά σιγά, αλλά είναι ανεπανόρθωτη η βλάβη. Πρέπει να μιλάτε πιο σιγά. Λοιπόν, ναι. Η, απουλία, η ΆΡΠΑ, μάλλον η αρχή αυτή της απουλίας, έκανε μελέτες. Βλέπει ότι υπάρχουν ακόμα την παρουσία της διοξίνης αλλά και μιας άλλης ουσίας γύρω εκεί στην περιοχή, ακριβώς γιατί είναι πάρα πολύ ε, ρυπασμένο το έδαφος. Ξεκολουθούμε όμως να περιμένουμε στοιχεία για τη δειγματοληψία. Δεν έχουμε καμία πληροφορία μέχρι στιγμής. Δεν έχει γίνει ουσιαστικά αυτή η έρευνα. Οι Ιταλικές αρχές δεν μας υποστηρίζουν. Βλέπουμε ότι το τάραντο σήμερα έχει πάρα πολύ μεγάλη ε, παρουσία νευρολογικών, καρδιογειακών παθήσεων, καρκίνων και άλλων νόσων. Και κοντά στην Ήλβα βλέπουμε ε, ένα στους 18 είναι καρκινοπαθής. Και όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στις εγκαταστάσεις, τόσο πιο μεγάλη είναι η συχνότητα αυτών των κρουσμάτων. Το Τάραντο έχει 200.000 περίπου κατοίκου. Διαβρέχεται δύο, δύο πλευρές από τη θάλασσα και η αλλιευτική δραστηριότητα ήταν η βασική δραστηριότητα πριν ε, την ανέργεια του εργοστασίου της Σίλβα και την ε, ιδιωτικοποίηση του 1995. Η κατάσταση ήταν ήδη δραματική, όμως ήδη το 2002 είχαμε στη Γένοβα, στο Κορνιλιάνο, ε, κάποια ε, μονάδες που μεταφέρθηκαν ε, στην περιοχή μας, γιατί δεν τα ήθελε η Γένοβα εκεί. Το 2005 πιστώθηκε ότι υπήρχε στον Τάραντο διοξίνη. Οι Ιταλικές αρχές δεν είχαν όμως δώσει τα σχετικά στοιχεία. Το 2008 ξεκίνησαν δύο ενώσεις να αναλύουν αυτόνομα τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το 2011 και τα προϊόντα αλίας ε, τέθηκαν ε, σε υποέλεγχο. Μιλάμε για μια τεράστια ε, μονάδα που έχει απαρχαιωμένες τεχνικές, παλιούς, παλιές μονάδες, δεν συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η ανάλυση που έγινε για τη συντροφική αλυσίδα έδειξε παντού την παρουσία διοξίνη, στα ψάρια, στα γαλακτοκομικά, στο ζωικό, στο κρέας κτλ πολύ μεγάλη μόλυνση από διοξινή, αλλά έχουμε και εκπομπές στην ατμόσφαιρα. Ε, κλείονται άλλοι ρήποι στην ατμόσφαιρα, στο τάρτο και αυτό επίσης δυσκολεύει τα πράγματα. Βενζόλιο, βενζοπυρίνιο, ε, φλωράνθρακες ε, και άλλες ουσίες. PCB λοιπά Και βέβαια ε, και ε, αναπνευστική, ε, αναπνευστικές γνώση έχουν προκληθεί. Δεν τα λέω εγώ, υπάρχουν επιστημονικές εκθέσεις και πρόσφατα είχαμε μια υψηλή σύμβαση με χιλιάδες σελίδες έγγραφα που υποστηρίζονται και από βίντεο και από εικόνες. Βλέπουμε ότι μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού έχει επηρεαστεί. Δεν είναι φυσιολογικά αυτά που συμβαίνουν στο Τάραντο. Αυτά που συμβαίνουν όμως ε, στο, χάρα, στο Τάραντο δεν θα μπορούσαν να συμβούν κάπου αλλού. Και ούτε με την ένοχη σιωπή των Ιταλικών αρχών που ήξεραν, αλλά δεν σταμάτησαν την παραγωγή της Ήλβα. Γιατί η Ήλβα είναι ένας εθνικός στρατηγικός πόρος για την Ιταλία. Το ξέραν οι αρχέ, το ξέραν από την αρχή. Προσποιούνται ότι δεν βλέπουν όμω, ακόμη και σήμερα. Και ουσιαστικά κάνουν ό,τι μπορούν ώστε η Ήλβα να συνεχίσει ε, την παραγωγή τη όπω συνέχισε τα τελευταία 20 χρόνια. Εγώ είμαι εδώ για να σα ε, μεταφέρω αυτή την κατάσταση, αυτή τη μαρτυρία, ότι η κατάσταση δεν έχει αλλάξει καθόλου στο τάραντο. Και όλα τα υποτιθέμενα μέτρα τα οποία έχουν λάβει οι φορεί οι αρμόδιοι δεν είναι αποτελεσματικά. Και αν ήταν αποτελεσματικά δεν εφαρμόζονται ούτως ή άλλως. Πεθαίνουμε από την μόλυνση, ε, από την ατμοσφαιρική ρήπαση, από τη διοξίνη. Μπορούμε να πεθάνουμε επειδή αναπνέουμε δηλητήριο, βεβαίως και μπορούμε. Ζητούμε τη βοήθειά σας. Σας ε, φέρω εδώ τις απεγνωσμένες ε, μαρτυρίες ε, γυναικών, μητέρων, που τα παιδιά τους χειρουργούνται για καρκίνο στα νοσοκομεία, τη φωνή των εργαζομένων που θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται χωρίς να χάσουν τη ζωή τους. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. η δικαιοσύνη δεν μας ε, ε, χορηγείται, δεν μας απονέμεται στη, στο τάρατο. Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες. Θέλουμε τη βοήθειά σας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Γιάν Κοντέσκου, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως ανέφερε η κυρία Μπατάλια, η Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία παράβασης κατά της Ιταλίας ε, στην περίπτωση αυτή. Μας ανησυχούν οι ανεξέλεγκτες εκπομπές ε, κατά την διαδικασία παραγωγής χάλιβα. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ε, παραβάσεις της οδηγίας IPPC. Αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη διαδικασία περιμένουμε την απάντηση των Ιταλικών αρχών υπάρχουν υποσχέσεις ότι κάτι κάνουν, λαμβάνοντας υπόψη όμως το επίπεδο ρήπανσης εκεί. Με βάση τα στοιχεία που μας έχουν υποβληθεί, θέλουμε να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα από τις Ιταλικές Αρχές και περιμένουμε την απάντησή τους μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου. Ευχαριστώ. Ζητάει κανείς άλλο το λόγο. Παρακαλώ. Θα ήθελα να γνωρίζω από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής γιατί σε μία ε, ε αναφορά που υπολήθηκε το 2007 έχει δοθεί απάντηση το 2010 και κατόπιν έχουν 2011 και μετά έχουν περάσει ε, πάλι δύο χρόνια και η Κομισιόν λέει ότι αναμένεται απάντηση. Εγώ θα ήθελα να ασκηθεί πίεση, να προχωρήσουν πιο γρήγορα τα πράγματα. Μπορεί η διαδικασία να προχωρεί καλά, αλλά ε, τη στιγμή που είναι τέτοια η κατάσταση δεν, μπορούμε να δεχτούμε τέτοιες καθυστερήσεις. Περιμένω από την Κομισιόν ε, να πιέσει τα πράγματα. The colleague the Βλέποντας τα δεδομένα αυτά και ακούγοντας την αναφορά, ε, την παρουσίαση κατάσταση από την αναφέρουσα και έχουμε και αυτή την αναφορά το 2007. Καταλαβαίνουμε το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και λόγω έλλειψης της δέωσης επιμέλεια από την Κομισιόν και γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγεία και γι' αυτό πιστεύω θα πρέπει να επιμείνουμε στην Επιτροπή μας. Η κατάσταση, μάλλον η δράση της ε, Ιταλικής κυβέρνησης ήταν να τα καλύψει τα πράγματα. Αφήνει τα πράγματα έτσι, δεν ε, εφαρμόζει τις ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως αυτή για τις εκπομπές, το 2010 ή περιβαλλοντική ευθύνη, οδηγία του 2004 και παρά το ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία επιβολής κυρώσεων το Σεπτέμβριο από την Κομισιόν κατά της Ιταλίας για να είμαστε μάλλον για λόγους προφύλαξης, πρόληψης και ξέροντας τους ρυθμούς με τους οποίους κινείται η Κομισιόν νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή ε, την αναφορά ακόμη. Να περιμένουμε να λυθεί το θέμα από την Κομισιόν γιατί οι Ιταλικές αρχές μετά από μια ολόκληρη σειρά παραλήψεων αθετήσεων ε, και με όλες αυτές τις προσπάθειες να συγκαλύψουν αυτό το θέμα, ε, δεν ξέρω τι ελπίδες έχουμε, ίσως ζητάμε πολλά, δεν ξέρω, μπορεί να μην περιμένουμε πολλά. No, okay. Please a colleague. Madam Chair, I'm not a... Δεν είμαι μέλος Τη επιτροπή αυτής, κυρία Πρόεδρε. Αλλά μπαίνω στον πειρασμό να πω και εγώ δύο λόγια, ενθαρρυντικά λόγια, προς τους συντάκτες αναφορά. Είναι σημαντικό, νομίζω, να υπάρξει μια, ένας απόϊχος, μια υποστήριξη, να αισθανθούν ότι τίνει ευήκονου στο Κοινοβούλιο για αυτά τα προβλήματα την τελευταία φορά που πήρα το λόγο σε αυτή την ε, επιτροπή μιλούσαμε για θέματα μόλυνσης ε, στη Βόρεια Ιταλία, στην Τεργέστη. Τώρα για... μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Έχω πάει στον Τάραντο, ε, ξέρω το πρόβλημα, ξέρω τις ανησυχίες του πληθυσμού, ξέρω το μέγεθος του προβλήματος, το οποίο είναι πολύ σοβαρό και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και μάλιστα γρήγορα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ουδής άλλος. Θα δώσω ένα λεπτό στην ε, συντάκτρια, αλλά μόνο ένα λεπτό για να απαντήσει. Ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό που μας απασχολεί πιο πολύ είναι το ότι θεωρούμε πως η Ιταλική κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει κάνει βήματα τα περασμένα χρόνια και να επιλύσει το πρόβλημα στον Τάραντα. Υπήρχε ένα περιβαλλοντικό σχέδιο ε, το οποίο δημοσιεύθηκε πριν από λίγες μέρες και που αφορούσε και την Ήλβα και που είναι μεγάλη ε, απογοήτευση για μας γιατί όλες οι επιταγές ε, ε, όλων των φορέων που θα έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί μέχρι το 2012 και 2013, τώρα ε, δεν εφαρμόζονται και έχει παραταθεί η προθεσμία για το 2015-2016. Μιλάμε για τα πιο σημαντικά βήματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για να ζήσουν οι άνθρωποι, ε, για να μπορούν οι κάτοικοι της περιοχής να αναπνέουν και να μην ασφικτιούν. Η Πρόεδρος, προφανώς πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή η προκύπτει αυτό σαφές, σαφέστατα και λόγω της ε, ανοιχτής διαδικασίας επί παραβάση. Θα ήθελα να πω στην Κομισιόν ότι ασχολούμαστε με αυτήν την αναφορά το 2007 και μετά από έξι χρόνια η Κομισιόν αποφάσισε να ξεκινήσει διαδικασία επί παραβάση. Μόνο μετά από έξι χρόνια. Όταν έχουμε να κάνουμε θέματα που αφορούν τη μόλυνση, αφορούν, αυτά τα θέματα, τα ίδια θέματα αφορούν την υγεία και τη ζωή. Έξι χρόνια τη χρειάστηκαν τη Επιτροπή για να αντιδράσει και είναι μια μεγάλη περίοδο. Δεν μπορεί ο κόσμο να περιμένει έξι χρόνια. Η έκκλησή μου είναι η Κομισιό να κάνει τη δουλειά της πιο γρήγορα. Πρέπει να επιταχύνει τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά. Γιατί οι κάτοικοι του Τάραντ δεν μπορούν να περιμένουν τόσο πολύ. Και αν μπορώ να κάνω και άλλη μια έκκληση στην Κομισιόν, θα ήταν η εξή. Να διορθώσει αυτά τα σημεία που θα κάνουμε και μάλιστα και μια επιστολή που θα την παρακαλούμε να, τα... να λάβει μέτρα. Το θέμα δεν είναι να εκκυρώνει μόνο, να τιμωρεί τις χώρες, να λαμβάνει μέτρα κυρωτικά. Το θέμα είναι να θεσπίζει και κάποιους στόχους. Και ο μείζον στόχος θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της ζωής των πολιτών, του περιβάλλοντος, αλλά και των θέσεων απασχόλησης και του παραγωγικού δυναμικού. Η Κομισιόν γιατί υπάρχει. Για να παρεμβαίνει συνολικά για όλα τα προβλήματα. Ελπίζω να το κάνετε αυτό. Με βάση τη διαθεσμική συμφωνία που έχουμε, η Κομισιόν πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή Αναφορών, ελπίζω να το κάνει, για τα μέτρα που θα λάβει και αν μπορεί να συμπεριλάβει και την Επιτροπή μας στις όλες προσπάθειες που θα κάνει, δηλαδή να την κρατάει ενήμερη και να την εμπλέξει στις προσπάθειες που θα κάνει. Θα κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά. Ευχαριστούμε τους ε, συντάκτες αναφοράς, τη συντάκτρια προκειμένου. Allora, adesso passiamo Πάμε στο σημείο 10. Πάμε στην ε, ψηφοφορία, στην εξέταση των τροπολογιών της έκθεσης για τη διερευνητική επίσκεψη στην Πολωνία. Μια στιγμή. I don't think so. Uh, wants to... Κύριε Μποστινάρου, θέλετε το λόγο. Όχι. Για τη Δανία. Για αυτό το σημείο θέλετε το λόγο. Όχι, μπορούμε να ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε την έκθεση αυτή. Πρώτον, τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ, κατά, αποχές, υποστηρίζεται. 2. Υπέρ, Η τροπολογία 2 έχει και προφορική τροπολογία ενσωματωμένη. Υπάρχουν αντιρρήσεις στην προφορική τροπολογία. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 2 με την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5. Με την προφορική τροπολογία. Αντιρρήσεις στην προφορική τροπολογία. Όχι. Ψηφίζουμε την 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7.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 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 19 καταπίπτει 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ με την προφορική τροπολογία αντιρρείς την προφορική τροπολογία όχι ψηφίζουμε την 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 α, αποσύρεται 22 τελική ψηφοφορία υπέρ κατά εγκρίνεται μόνο με δύο ψήφους κατά Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στη δεύτερη έκθεση. Κυρία Βέρτμαν, θέλετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας παρακαλέσω να δείξετε λίγη υπομονή, γιατί γίνανε κάποια περίεργα ε, ενδιαφέροντα πράγματα σε διαφορετικές τροπολογίες και τα συμπεράσματα το Αν θυμάστε, στο γραφείο του Δημοσολαβητή κάναμε μια συνάντηση απουσία του, εκπροσωπήθηκε από κάποια μέλη ε, του γραφείου του. Η έκθεση μιας διερευνητικής επίσκεψης μπορεί μόνο να επαναλαμβάνει αυτά που ελέγχθησαν, έγιναν, που υπόθηκαν, που είδαμε, που ακούσαμε. Στις 3 Οκτωβρίου ήρθε επαφή μαζί με το γραφείο ενός συναδέλφου και συγκεκριμένα το γραφείο του Δανέζου διαμεσολαβητή ήθελε να αλλάξουν κάποια κομμάτια της έκθεσής μας. Φυσικά, ε, όπως και εξπακούεται, έθεσα το θέμα υπόψη ε, της αντιπροσωπείας μου και όλοι μας ε, είπαμε και συμφωνήσαμε ότι δεν μπορεί να αλλάξει η έκθεση δεν θέλουμε να αλλάξει έκθεση ε, και να περιλαμβάνει πράγματα που δεν υπόθηκαν, που δεν συζητήθηκαν. Αυτό θέλω να το θέσω υπόψη σας, διότι όλοι πρέπει να το ξέρετε, πιστεύω. Ενημέρωσα ε, και τη συνάδελφη με το ίδιο μα λέγοντας ότι δεν το κάνει με αυτό που μας ζητεί το. Εμείς μπορούμε να καταγράφουμε μόνο όσα ήδη έχουν γίνει στην πράξη. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Όχι μόνο προς τους συναδέλφους. Όλοι πρέπει να γνωρίζουν τι γίνεται παρασκηνιακά. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον κατάλογο ψηφοφορίας τώρα. Σας εξηγώ εν συντομία ότι υπήρξαν κάποιες τροπολίες από συνάδελφους που δεν ήταν μέσα προσωπίας, Κάποιες είναι καλές αλλά δεν αντικατοπτρίζουν την κατάσταση, δεν εμπίπτουν στο παιδί της Αποφασίσαμε λοιπόν να έχουμε αρνητικό πρόσημο οι τρεις ε, βουλευτές που είμαστε μέσα της Επίσης δεν μας άρεσε η κατάσταση. Υπάρχει μια τροπολογία που δεν μας ικανοποιεί. I would like to request, please, uh, that... Και γι' αυτό θα βάλουμε αρνητικό ε, πρόσημο. σε ό,τι δεν αφορά ε, το ότι μας προσέγγισαν και μας ζητήθηκε να αλλάξουμε ε, την έκθεση, θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Βέρτμα. Θέλατε για τη διαδικασία το λόγο. Θέλω να διαβάσω κάτι που έγραψε η Μάργκρετ Άουκεν. Μα δεν είμαστε τώρα στη συζήτηση, λέει πρόεδρο, είμαστε ψηφοφόροι. Ναι, αλλά μου έστειλε η κυρία Άουκεν για την ψηφοφορία τη θέση τη. Μπορώ να τη διαβάσω. Για την κυρία Άουκεν, ναι, μάλιστα. Όχι, μισό λεπτό, λέει πρόεδρο. Δεν είναι συντάκτρια η κυρία Άουκεν. αν θέλετε μας δίνετε αυτό το έγγραφο να το λάβουμε στα πρακτικά ε, υπόψη, να το συμπεριλάβουμε στα πρακτικά. Να διαβάσετε τώρα το κείμενο όχι. We open the vote. Ε, Ξεκινάει λοιπόν η ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Α, η, 5, η 4 καταπίπτει. Πάμε στην 5. Τροπολογία 5 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 6 ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Πού πάει αυτή η προφορική τροπολογία? στην έκτη σύσταση υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Υπάρχει αντίρρηση. Όχι. Άρα ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπέπτει επόμενη. Πάμε στην 9. πέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. 11 γιατί 10 καταπίπτει. Υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχέ. εγκρίνεται. Συμβεβαστική τροπολογία στην 11η σύσταση 11α νέο. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Α, ε, κατά. Αποχές. Να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. 18 ψήφι υπέρ. Μπορείτε να συμφωνήσετε μεταξύ σας. Λοιπόν, ποιος είναι υπέρ της Τροπολής 18. 5. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 προς 5. Δεν υπήρχαν αποχές. Άρα ερχόμαστε στην τελική ψηφοφορία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η έκθεση. Με μία ψήφο κατά. Ευχαριστώ όλες και όλους. Και τους συντάκτες. Συνάδελφοι, πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε την έκθεση για την Ελλάδα. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Τουργκάη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος γιατί είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλους και ιδίως όσους με συνόδευσαν στην αποστολή αυτή. Τον Μάριο Μπαλντίνη, μάλλον Μαρίνο Μπαλντίνη που είναι εδώ, και από τον συνάδελφο της, Επιτρο... της ομάδας των Πρασίνων, τον κύριο Γκούντι. speaking. Μιλάει ο κύριο Ετουργκάιθ, παρακαλώ. Ακούστε τον. Σα ευχαριστώ κύριε Πατρά. Έλεγα λοιπόν ότι θέλω να ευχαριστήσω του ε, συνάδελφου που με ε, συνόδευαν, αλλά να ευχαριστήσω και την ε, κυρία Παλιαδέλη, τον κύριο Χουντή και τον κύριο Σαλαβράκο που ήταν τα λεγόμενα εξοφίκιο μέλη από την Ελλάδα δεν ήταν μόνο μια αποστολή που θα έχει ως αποτέλεσμα την εκπόνηση έκθεσης από τον συνάδελφο από την Κροατία ή τη Γερμανία ή εμένα, αλλά μια έκθεση που θέλουμε όλοι να την προσυπογράψουν, και οι Έλληνες ε, και όσοι δεν είμαστε Έλληνες. Ήταν εξαιρετική η επίσκεψη. Να ευχαριστώ τη γραμματεία, ιδίω την ε, Ναταλία, και γιατί μου έφερε και ένα χάπιο τον πονοκέφαλο, αλλά και γιατί με βοήθησε, μας βοήθησε. Και πριν πάμε στην Ελλάδα, μας ενημέρωσε με ένα έγγραφο υποδειγματικό. Δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο. Γιατί έχω ξαναπάει ε, σε άλλες δερματικές αποστολές, δεν έχω ξαναδεί τέτοια δουλειά. Πάρα πολύ καλό το κείμενο το ενημερωτικό ε, και αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, είχαμε διάφορες επαφές και ήταν πάρα πολύ επιτυχημένες και η στήριξη που είχαμε από τις ελληνικές αρχές. Και η στήριξη που είχαμε από τους αναφέροντες έκαναν πολύ εύκολη την αποστολή μας και πρέπει να σας πω ότι δεν υπήρξε καμία δυσκολία, καμία τριβή, κανένα πρόβλημα. Το αντίθετο ε, ήταν ε, πολλές οι πάρα πολύ θετικά κύλησαν όλα. Βέβαια ήταν πολύ πλοκή η αποστολή μας, γιατί ξέρετε ότι είχαμε να πάμε σε πολλές ε, περιοχές που απήχαν μια από την άλλη. πήγαμε στην Αθήνα, στο Γραμματικό, στην Πελοπόννησο, στην Κέρκυρα και στη Βορρά Ελλάδα. Στα αλβανικά σύνορα κοντά. Επιμένω ε, και επαναλαμβάνω ότι μας έκαναν, ε, μάλλον μας ε, πάρα πολύ εύκολη την επίσκεψη και όσοι ήταν εκεί, οι αναφέρτες μας εξήγησαν τους στόχους, και είδαμε επιτόπου ό,τι θέλαμε. Όλα όσα ζητήσαμε τα είδαμε. Το λέω ξεκάθαρα αυτό. Δεν είχαμε ένα πρόβλημα. Είχαμε πρόσβαση ε, σε, στις ε, χωματερές και με όλους όσους θέλαμε να συναντηθούμε, με υπαλλήλου των δημαρχείων, με την κυβέρνηση, όλα ήταν ε, δυνατό να γίνουν χωρίς πρόβλημα. Όπως σας προείπα κυρία Πρόεδρε, αυτή είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων είναι εδώ ο συνάδελφος που ήταν μαζί στην επίσκεψη, δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι. Από εκεί και πέρα τώρα. Θα καταθέσουμε τροπολογίες. Θα έχω σύντομα την, ε, το σχέδιο της έκθεσης έτοιμο στο διανύμο. Και γι' αυτό θέλω να ολοκληρώσω εδώ ευχαριστώ για μία ακόμη φορά τη γραμματεία, τον Ντέιβιτ που ήρθε μαζί. Αλλά μου επιτρέψατε, Ντέιβιτ, ε, ελπίζω χωρίς πρόβλημα. Ε, θα ήθελα να αναφέρω και τις δύο Ελληνίδες ε, που ήταν εκεί και τους συναδέλφους μου, τους δύο βουλευτές που ήρθαν μαζί μας. Είμαστε διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση τυχόν έχετε. Παραλαμβάνω ότι σύντομα θα έχετε στη διάθεσή σας την έκθεσή μου, οπότε θα μπορούμε να ε, συζητήσουμε πάνω στο κείμενο πια. Κύριος Μποργκίνη. αν, μου επιτρέπετε, ε, μια και δεν υπάρχει μετάφραση από τα κροατικά, ας μιλήσω ιταλικά. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε ο προλαλής σας. Σε αυτή την αποστολή στην Ελλάδα ε, όντως ε, είχαμε τα πράγματα κύλησαν όπως τα είπε, αλλά ξέχασε ίσως ε, να πει κάποια πράγματα τα οποία ήταν λίγο αρνητικά ε, χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε διαδηλώσεις. Ε, Παρ' όλα αυτά, χάρη στην καλή οργάνωση, όλα πήγαν κατευχήν στο τέλος. Ενημερωθήκαμε από όλου. Μας έδωσαν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία, όλες οι αρχές, όχι μόνο οι συντάκτες, αλλά και οι αρχές, οι υπουργοί, οι περιφερειακές αρχές, οι περιφερειάρχες, δηλαδή οι δήμαρχοι, τα πανεπιστήμια, το, καπα, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με... είχε όλα τα στοιχεία τα ενημερωτικά στη διάθεσή μας και οι πολίτες και οι εκπρόσωποι των κομμάτων όλοι μας βοήθησαν για να ενημερωθούμε. Νομίζω ότι πραγματικά ενημερωθήκαμε θαυμάσια, απρόσκοπτα. Ήταν για μένα η πρώτη αποστολή που έκανα στην Ελλάδα. Είμαι καινούριο μέλος στο Ευρωκοινοβούλιο. Είμαι Κροάτης και έγινα Ευρωβουλευτής από 1η Ιουλίου. Και πραγματικά εντυπωσιάστηκα από τον τρόπο που δουλεύουν στην Ελλάδα, χωρίς καθόλου διαλύματα. Ξεκινάνε να δουλεύουν πάρα πολύ νωρί το πρωί και δουλεύουν μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Και δεν κάνουν καν διάλειμμα για φαγητό. Οργάνωσαν δε πάρα πολύ ωραία τι μετακινήσει που ήταν πολύ άριθμε. Δουλέψαμε πάρα πολύ, αλλά νομίζω και καλά. Υπήρχε απόλυτη ενημέρωση οι, όλοι οι αρμόδιοι ήταν παρόντες, νομίζω ότι πραγματικά έγινε μια θαυμάσια δουλειά. Eh, eh, eh, Δεν θέλει άλλο το λόγο, οπότε θέλω και εγώ να ευχαριστήσω ξανά το προσωπικό, τον Ντέιβιτ, τον Αντών, τον Μάρκ, τους ε, υπαλλήλους από τις ομάδες που ήρθαν μαζί μας. Ε, ζητώ συγγνώμη γιατί σας ξέχασα πριν, αλλά ήθελα να σας ευχαριστήσω και εσάς για την παρουσία σας, για τη στήριξή σας, ε, τη βοήθειά σας. Και στις επόμενες, πώς να το πω, ναι, συνεδριάσεις σε Επιτροπής Αναφορών, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να συζητάμε το θέμα αυτό, έχοντας πλέον τα έγγραφα στη διάθεσή μας. Και βέβαια θα ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία με την ε, ψηφοφορία του εγγράφου αυτού. Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά όλες και όλους. Ο, η Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και με αυτό το σημείο της μέρης διάταξη. Τώρα λοιπόν διακόπτουμε τις εργασίες της Επιτροπής και περνάμε στις συνεδρίες των συντονιστών. Έγινε μια πρώτη συζήτηση. Θα επανέλθουμε για την ε, επίσκεψη στην Ελλάδα σε μια προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Περνάμε στην συνεδρίαση των συντονιστών.